Θα επαναλάβουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτύξεως και αυτή τη φορά το θέμα είναι οι συνέπειες της, ε, ε οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης επί των αναπτυσσομένων χωρών. ønsker deg hjertelig velkommen. I'm also very happy to... Συνεχίζει στα αγγλικά η πρόεδρος μετά από ένα σύντομο διάλειμμα στα σουηδικά. Θα ήθελα να απευθύνω το καλώς ορίσατε στην Αμινάτα Τραόρε, ε, συγγραφέα από το, Μαολί, από το Μάλι. Έχει διατελέσει υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού στο Μαλί και είναι και πρώην συντονίστρια του ε, Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και είναι και η τρέχουσα συντονίστρια για ε, τρέχοντα θέματα για εξωτερικής πολιτικής του Μαλή. Επίσης είναι και γνωστή επικρίτρια της παγκοσμιοποίησης. Ε, επίσης κοντά μας είναι ο κ. Μαρκ Πλάντ του IMF. αρμόδιος για την Αφρική και πρώην υπεύθυνο για την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις σχέσεις με τις φτωχότερες χώρες. Και όπως είπα στην αρχή είμαι προσωπικά πολύ ε, χαρούμενη που μπορώ να υποδεχθώ τον ε, ε, νορβηγό εκπρόσωπο στην ακροασή μας, τον καθηγητή Σέλντρεκ, ο οποίος ε, ήταν και επικεφαλής Νορβη, ε, Επιτροπής Νορβηγικής Κυβέρνησης για τα, τις παράνομες ροές ε, κεφαλαίων χρημάτων. Στην παρουσίασή του θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις, παράνομε παράνομες εκροές χρημάτων από αναπτυσσόμενες χώρες. Κοντά μας είναι και ο κύριος Ρέιμον Μπέικερ, διευθυντής και επισκέπτης καθηγητής στο Brooks Institute. Έχει συγγράψει το βιβλίο «Η αχίλιος πτέρνα του καπιταλισμού, το βρώμικο χρήμα και πώς ε, μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση». Ειδικό για θέματα πλησίματος ε, του βρώμικου χρήματος και άλλα σχετικά, καθώς και τις συνέπειες των ε, δράσεων αυτών στις διοικητικές οικονομίες. Εν τέλει, Κοντά μας είναι ο κύριος Πέτρο Ντεβασκονσέλος, συντονιστής της IFAD, Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα μιλήσει για την σημασία των εμβασμάτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Προέρχεται από το G20, έρχεται μάλλον από το G20 όπου μόλις παρουσίασε την ε, παρέμβασή του και μεγάλη ικανοποίηση τον υποδεχόμαστε σήμερα. Θα δώσω τώρα την διεύθυνση της συζητήσεως στον συνάδελφό μου κύριο Γκερέρο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είπα και πριν ότι η ε, πραγματική και φυσική πρόεδρος μας είστε εσείς. Εγώ απλώς θα διευθύνω την συζήτηση ε, αφού μάλλον πρώτα ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας και αφού ευχαριστήσω και όλες και όλους εσάς που είστε εδώ θα συντάξουμε έκθεση για τις συνέπειες ε, της χρηματικής, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Πλάντ για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Σας εύχομαι ε, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να απευθύνω λίγα λόγια στην Επιτροπή σας ε, εξ του IMF. Το IMF ε, ανισχύει ιδιαίτερα για την παγκόσμια οικονομική κρίση, την χειρότερη ε, παγκόσμια οικονομική κρίση από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η οποία απειλεί να σπρώξει στη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους. 8 έως 10 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να πέσουν στη φτώχεια εάν η διεθνή κοινότητα δεν αντιδράσει και γρήγορα. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Το IMF είναι, παίζει ηγετικό ρόλο στον κόσμο ε, για να, και ε, προειδοποιεί σχετικά με τι συνέπειε. Έχουμε ήδη προσφέρει συμβουλέ στι ε, χώρε μέλη μα για το πώ να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ζητήσαμε αύξηση πιστώσεων κυρίως υπέρ των πιο ευάλωτων ομάδων και σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Και έχουμε προσφέρει και δανειοδοτήσεις ακόμα πιο ε, φθηνέ. Θα έρθω σήμερα στην ε, υποσαχαρική Αφρική. Αλλά πολλά εξ όσων θα πω ισχύουν και για πολλές άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Πρώτα, οι οικονομικές αναταραχές που πέρασε η Αφρική ε, πρόσφατα. Μεταξύ 2002 και 2007 η αύξηση του εισοδήματος της παραγωγής μάλλον στην Αφρική ήταν 6,5%. Ο πληθωρισμός είχε πέσει σε, χαμηλό επίπεδα, σε χαμηλά επίπεδα σε όλες σχεδόν τις χώρες. Μετά όμως η Αφρική επλήγει από δύο ε, σημαντικά σοκ. Πρώτον, η αύξηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων ε, στις αρχές, στο 2007 και 2008 προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις κυβερνήσεις. Και αργότερα, το 2008, άρχισε η μεγάλη ύφεση με προϋπολογισμούς οι οποίοι ήδη αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και ε, τροφίμων. Τώρα αντιμετωπίζει η Αφρική και σημαντική μείωση των εξαγωγών της, σημαντική μείωση των εμβασμάτων των μεταναστών της και μειωμένη εξωτερική βοήθεια. Οι ε, εκροές από την Αφρική αναμένεται να αυξηθούν μόλις κατά 1%. Για πρώτη φορά σε μία δεκαετία θα δούμε το κατακεφαλήν εισόδημα στην Αφρική να μειώνεται. Ε, κρίση έπληξε δυσανάλογα τις χώρες. Αρχικά περισσότερο χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία όπως η Νότια Αφρική. Επίσης οι χώρες οι οποίες βασίζονται σε ένα βασικά εξαγωγικό προϊόν όπως ε, το, ε, ο καφές ή το κακάο ή το πετρέλαιο ή το καουτσούκ επλήγησαν επίσης βαρύτατα. Συνέχισε όσο συνεχιζόταν η ε, ανάπτυξη της γεωργίας τα πράγματα πήγαιναν καλά αλλά σε όλη την Αφρική υπάρχουν σημαντικές ευάλωτες ομάδες, σημαντικές ε, ε, σε αριθμό δηλαδή. Πώς ανταποκρίνονται τώρα οι αφρικανικές χώρες στην κρίση. Μια πρόχειρη απάντηση είναι ότι τα καταφέρουν καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Σε παλαιότερες κρίσεις είχαν πολύ περιορισμένο περιθώριο λιγμών για να αντιμετωπίσουν τέτοιες υφέσεις. Είχαν μεγάλα κενά στους προπολογισμού, σημαντικά χρέη και ήταν πολύ ευάλωτες οι χώρες απέναντι σε παλαιότερες κρίσεις. Δεν είχαν αποταμιεύσεις και επομένως δεν είχαν κανένα περιθώριο. Ήταν υποχρεωμένες να κάνουν περιοριστικές πολιτικές, να επιβάλλουν εξαιρετικές, ε, εξαιρετική λιτότητα. Βεβαίως αυτές ήταν λανθασμένε απαντήσει αυτέ. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βρισκόντουσαν σε καλύτερη θέση στην αρχή τη ύφεση. Για το σύνολο τη περιοχή αυτή, για το 2007 και 2008, οι ε, χώρε αυτέ είχαν ήδη κάποια μέτρια πλεονάσματα στου προπολογισμού του. Και έχουν αναλυθεί και πρωτοβουλίε άφηση του χρέου, οι οποίε ε, συνέβαλαν πολύ σε μια καλύτερη θέση των χωρών. Είχαν λοιπόν κάποιες οικονομίες οι χώρες κάποια αποθέματα. Ήταν λοιπόν σε ευνοϊκότερη θέση αφετηρίας. Τους προσέφερε κάποια περιθώρια ελιγμών. Αυτά τα περιθώρια ελιγμών πολλές από τις χώρες της Αφρικής τώρα τα χρησιμοποιούν. Θα αυξηθούν σε τρεις από, τέσ, από τις τέσσερις ε, ευρωπαϊκές, σε τρεις από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες θα αυξηθεί ε, το έλλειμμα του ε, ισολογισμού. Πάντως κατάφεραν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Ορισμένες χώρες όπως η Μποτσουάνα ή η Τανζανία έχουν μάλιστα αυξήσει τις ε, ε, δαπάνες τους κάνοντας αντικυκλικές κινήσεις. Έχει ενισχυθεί και η βοήθεια απ' έξω για τις χώρες αυτές. Ευτυχώς ο κίνδυνος του πληθωρισμού παραμένει μέτριος. Έτσι μπόρεσαν ορισμένες χώρες να ε, χρησιμοποιήσουν τα ε, επιτόκια λιγότερο ως ε, περιοριστικό παράγοντα για την αύξηση του πληθωρισμού. Είμαστε λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 2010 και για μια ενδεχόμενη ανάκαμψη για τις χώρες της υποσαχαρικής Αφρικής. Η πρόβλεψή μας για την αύξηση του προϊόντος τους δια του χρόνου είναι περίπου 4%. Υπάρχουν όμως και σημαντικοί κίνδυνοι. Αν δηλαδή η παγκόσμια ανάκαμψη δεν υλοποιηθεί εν τέλει ή αν οι δωρητέ δεν προσφέρουν αρπαρκή υποστήριξη. Άρα χρειάζεται εποπτεία, παρακολούθηση και από τις κυβερνήσεις στην Αφρική και από τους εταίρους τους. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα επανέλθουμε στα επίπεδα πριν από την κρίση. Η ανάκαμψη και βασισμένοι ιδίω στα εμβάσματα και σε άλλους παραδοσιακούς παράγοντες δεν φαίνεται πιθανή. Μέτρα για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, να βελτιωθούν οι κεφαλαιαγορές, αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουν κρίσιμο χαρακτήρα. Οι προσπάθειες αυτές θα χρειαστούν σημαντική ενίσχυση από τη διεθνή κοινότητα και για πολλά χρόνια μετά από την, από το ξεπέρασμα της κρίσης. Πώς αντιμετωπίζει τώρα το IMF ε, την κρίση στην Αφρική και σε άλλες ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Αυξήσαμε πρώτα τις πιστώσεις που δίνουμε στην Αφρική. Αυξήσαμε ε, σημαντικά τη χρηματοδότηση προς χώρες χαμηλού εισοδήματος από πέρσι, από τον Σεπτέμβριο. Φτάσαμε να δίνουμε δανειοδότηση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το 1,1 δισεκατομμύριο ε, για το ε, ολόκληρο το 2008 και ε, σχεδιάζουμε ακόμα περισσότερα μέτρα. Μέχρι το 2014 θα αυξήσουμε τα δάνεια που δίνουμε σε 17 δισεκατομμύρια και πολλά αυτά με προκαταβολές για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάνουμε επίσης τη δανειοδότησή μας πιο φθηνή, ακόμη και με μηδενικά επιτόκια και στο μέλλον γενικά τα επιτοκιά μας θα είναι χαμηλότερα. Έχουμε προσφέρει επίσης ε, χρηματοδοτήσεις με ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα. Οι χώρες της υποσαχαρικής Αφρικής έλαβαν ήδη ποσά του ύψους των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων που τους επέτρεψαν έτσι να ενισχύσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα για να έχουν και μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για το μέλλον, το οποίο ήδη χρησιμοποιούν από τώρα κάποια από τα περιθώρια αυτά ελιγμών. Αλλάζουμε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις δανειοδοτήσεις. Αντιλαμβάνομαστε ότι οι διάφορες χώρες έχουν διάφορες ανάγκες και άρα προσφέρουμε μέτρα κομμένα και <clears throat> προσφέρουμε ε, ενίσχυση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Αναλόγως με το αν οι ανάγκες είναι πολύ βραχυπρόθεσμες ή ε, πιο μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες. Κάναμε και αλλαγές στους όρους που επιβάλλουμε για την δανειοδότηση. Ορισμένα από τα δάνεια όπως αυτά της ταχείας αντίδρασης στην πραγματικότητα είναι, στην ουσία είναι μάλλον άνευ όρων και άλλα έχουν ε, γίνει, έχουν γίνει ιδιαίτερα λιτές οι διαδικασίες ώστε να ε, αντιμετωπίζονται καλύτερα οι ανάγκες. Εξακολουθούμε ε, να συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις, παρόλα αυτά δεν αναστέλουμε τις ε, εκταμιεύσεις από μέρους μας εάν δεν ανταποκριθούν σε όλα τα μέτρα που απαιτούμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα προγράμματα που ε, ε, ενισχύουμε ενισχύουν και συγκεκριμένους στόχους αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Στο Μπουρούντι ενισχύουμε την διανομή λιπασμάτων, τις μικροπιστώσεις και τη διατροφή στα σχολεία στην Γκάνα κοινωνικά προγράμματα για την ε, υγεία καθώς και, ε, και δωρεάν ε, τετράδια για τα σχολεία και έχω και πολλά άλλα παραδείγματα. Μια άλλη προσέγγιση είναι μια πιο εύκαμπτη προσέγγιση απέναντι στο χρέος. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες χαμηλής ανάπτυξης δεν έχουν επαρκή υποδομή για ανάπτυξη. Στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα μόνο να δίνουμε υψηλών επιτοκίων επιδοτήσει, Ε, μάλλον, ενώ γνωρίζουμε τώρα ότι έχουν σημαντικέ ανάγκες. Τώρα ε, οι χώρες αυτές θα μπορούν να δανείζονται περισσότερο και με concessional και με non-concessional loans. Αυτές οι προσπάθειες που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να βοηθήσει τι χώρε με επικοδομητικό τρόπο να ξεπεράσουν την κρίση και, τα, και τις της εξετάζοντας και τις ε, προοπτικές για μέσο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Τι θεωρούμε ότι χρειάζεται να κάνει η διεθνής κοινότητα. Πολλές από τις χώρες αυτές θα εξακολουθήσουν να παραμένουν εξαρτημένες σε σημαντικό βαθμό από εξωτερικές ροές κεφαλαίων και από τα διεθνή εμβάσματα. Επομένω, η υποστήριξη των διεθνών οργανισμών θα παραμείνει κρίσιμη. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή. Η χώρες αυτές θα χρειαστούν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια έξτρα χρηματοδότηση για φέτος. Πέραν των όσων ήδη τους υποσχεθήκαμε στην διάσκεψη κορυφής του Glenn Eagle πριν από δύο χρόνια. Και άλλοι διεθνείς οργανισμοί συμβάλλουν, αλλά όλοι οι δωρητές οφείλουν να παίξουν τον ρόλο τους με τρόπο συγκεκριμένο και ε, ζωηρό. Συνοψίζω σε τρία σημεία. Πρώτα, το IMF από την αρχή αντιλήφθηκε ότι η ε, παρούσα κρίση θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες χαμηλού εισοδήματο και θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους της χιλιετίας και ιδίως την μείωση της φτώχειας. Την ώρα που είχε αρχίσει να υπάρχει μια κίνηση προς τα εμπρός, έπληξαν την κρίση δύο σημαντικά σοκ. Οι πολιτικοί μας, οι συμβουλές μας είναι ξεκάθαρες ο αγώνα για την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία πρέπει να συνεχιστεί για την μείωση τη στόχιας. Άρα σε πολλέ χώρε θα χρειαστεί να χαλαρώσουν οι στόχοι για την ε, ισοσκέλιση των προπολογισμών και άλλων σε ορισμένε από τι ε, χώρε χαμηλότερου ε, εισοδήματο. Θα πρέπει τα αποθέματα που έχουν να τα χρησιμοποιήσουν. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη. Ήδη το IMF έχει αυξήσει τα ε, ποσά των δανείων και έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο κάνει δανειοδοτήσει. Δεν αρκούν αυτά. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να κάνει σημαντική προσπάθεια για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και τώρα, δώσουμε το λόγο στην κυρία Τραωρέ. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ και λαμβάνω μέρος σε αυτή τη ε, διαδικασία της αξιολόγησης των συνεπειών της κρίσεως. Από πλευράς αυτών των ε, φτωχών χωρών και πιο συγκεκριμένα της Αφρικής. Θα ήθελα τώρα να σας ε, αναφέρω ότι έχουμε μπροστά μας μια συστημική κρίση. Έχουμε εξαφάνιση, κατακρύμνηση των ε, κερδών, κάτι το οποίο βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ πιο οξύ ως πρόβλημα στην Αφρική, όπως είπε ο Προσταλής σας. Και έχουμε και κάποιες άλλες κρίσεις, ε, όμως που σοβούν χωρίς να έχουν τύχει τις ίδιες προσοχές και όπως θα μας κρίση στην ανάπτυξη. Και όσον αφορά την δημοκρατία. Πριν επομένως καταρρεύσει το σύστημα, είχαμε εκδήλωση της ε, κρίσης. Ήταν στα μάτια μας μπροστά. Λόγω της κρίσης που σοβούσε στις πρώτες ύλες. Επίσης όσον αφορά τα, τα προβλήματα τη προσαρμογή της προσαρμογής στην οικονομική αναδιάρθρωση γιατί είχαμε ε, πρόβλημα και ανεργίας αλλά και ε, μισθών πείνας που έπαιρναν πάρα πολλοί εργαζόμενοι ε, οπότε είχαμε πρόβλημα και κατά συνέπεια στην διατροφή είχαμε και οικολογική κρίση ξηρασία, μόλυνση, απερίμωση είχαμε επίσης και κοινωνική κρίση κατάρρευση του παλιού συστήματο τη Ελληνική και κοινωνική πρόνοια. κρίση ταυτότητας, συγκρούσεις, έλλειψη, σημείων που φτάνουν στον προσανατολισμό, οροσίμων, διαφθορά και ταυτόχρονα τιμωρησία. Και από όλε αυτές τις κρίσεις η χειρότερη, η πιο ανησυχητική είναι το ότι υπάρχει αιμονή σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ανάπτυξη. Που αυτό δημιούργησε αυτό το γενικευμένο χάο. Γιατί πρόκειται για μια χαοτική κατάσταση. Και δυστυχώ φτάσαμε σε τέτοιο σημείο που είχαμε πρόοδο ω 6% του ρυθμού ανάπτυξη για το οποίο κομπάζουν οι ηγέτες. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνει η νοικοκυρά στο καλάθι της ούτε οι έγκυες γυναίκες που χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας και αυτές που χρειάζονται φάει για τα παιδιά τους. Ούτε φαίνεται αυτό σαν οικονομικές ευκαιρίες που να μπορούν να μας βοηθήσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Και έρχονται λοιπόν ένα σωρό άνθρωποι και πνίγονται εδώ στις πύλες Ευρώπης. Οπότε τι θα πρέπει να γίνει με αυτή την κρίση, τι θα γίνει όσον αφορά τους πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει αυτές να αυξηθούν και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που ήδη είχαν οι κρίσεις χωρίς να μπορούν να έχουν βρει τις απαντήσεις. Είδαμε ότι ήταν να βρεθεί αυτό το, το λίγο χρήμα χρειαζόταν για να μπορέσουμε να τον αυτή την διατροφική κρίση, η οποία οδήγησε σε ένα δισεκατομμύριο κόσμο ο οποίο χτυπήθηκε από την τραπεζική κρίση και βλέπουμε πόσοι στην Ευρώπη έχουν εμπλακεί από αυτή την νοοτροπία των χρόνων της Βορείου Ευρώπης που ήταν αυτοί οι οποίοι επίκησαν την Αφρική. Την εκμεταλλεύτηκαν. Έχουν παράπονα τώρα οι Βόρειοι από τις τράπεζές τους. Όμως και εμείς έχουμε τα ίδια παράπονα από το Διεθνή Νομισματικό Ταμείο. Οπότε έχουμε αυτό το κλίμα και βρισκόμαστε σε, σε, ένα, σε ένα πλαίσιο όπου ποτέ δεν μπορεί κανεί να κάνει για όλα αυτά τα λάθη που ουσιαστικά είναι οικονομικά εγκλήματα στην Αφρική. Ουδέποτε συνειδητοποιήθηκε το γιατί και το πώ. Οπότε, ε, σε, κάποια στιγμή πήγαμε για απορριθμίσει, γίναμε για ιδιωτικοποιήσει, πήγαμε για πιέσει που ασκήθηκαν στα κέντρα απόφαση στην Αφρική. Όμω, αυτό ήταν η κρίση στη δημοκρατία. Άρα αυτό που σας λέω, σας τα λέω μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, τόσο ώστε να δείτε. Αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι μια διαδικασία που εντάσσεται ακριβώς στην, στον εορτασμό της πτώσης του τείχους. Γιατί έτσι μπήκε ένα τέρμα στις δικτατορίες και περάσαμε σε εκδημοκρατισμού, σε εκλογέ, ούτω ώστε ό,τι ανάπτυξη δεν ήταν την άλλη πριν χώρο να γινόταν τώρα. Ακριβώ γιατί έτσι είπαμε θα μπορούν να ελέγξουμε του άρχοντε. Όμω αυτό δεν γίνεται. Δείτε τι έγινε στην Γουινέα, τι σφαγέ έγιναν και είδαμε πόσοι δεσμοί γυναικών έγιναν και όλα αυτά καταλήγουν σε αυτή την εξάρτηση τέτοιου είδους ανάπτυξη που ελέγχεται τι πολυεθνικέ και εκμεταλλεύεται τι πρώτες ύλε. Άρα είμαστε είδο η διακινδύνευση διότι τώρα που σας μιλάω η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Αφρικανών δεν ξέρουν ποια είναι η αιτία της. Κανείς στην Αφρική δεν μιλάει για κρίση. Γιατί εκεί η κρίση είναι καθημερινή, συνεχής. Δημιουργήθηκε στη Δύση αυτή η κατάσταση και σήμερα υποχρεώνει το μέτωπο της κοινής γνώμης και της ε, ε, ηγετικής τάξης να μην μπορούν να αποφύγουν αυτή την κατάσταση και έτσι όμως τα πληρώνουμε εμείς ενώ μας λένε ταυτόχρονα ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην χαθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα, ό,τι κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια. Όμω, ποιο οφείλεται από αυτό, λέω. Για, με αυτό το ρυθμό που τρέχει η ανάπτυξη, ε, από ορυκτά, από τουρισμό, από πετρέλαιο, ό,τι ό,τι βγήκε, ε, δεν το καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσει κανείς ταυτόχρονα και την κρίση και αυτό το οποίο έγινε τα τελευταία 20 χρόνια. Την αποτυχία περισσότερο εκδημοκρατισμού. Και έτσι να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι η Φουκαριάρα, η Αφρική, ο μεγάλος χαμένος της παγκοσμιοποίησης, τα χρεωμένα κράτη της Αφρικής. Όμως εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι πρόκειται για την περιοχή του κόσμου που Μπορεί κανείς να δει μέχρι ποιο σημείο και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο που καταστρέφει το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο. Είναι η απόδειξη η Αφρική. Είναι το υπομόχλιο του ώστε να μπορέσει κανείς να βγει από την κρίση. Την κρίση την οποία την, την κοιτάμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. εμένα δεν με συγκινεί η ιδέα τη αναδυόμενη ε, οικονομία, γιατί ξέρω που καταλήγει αυτό. Αυτό που με ανησυχεί είναι αυτή η ταπεινωτική κατάσταση. Αυτή η συγκατάθεση, συγκατάβαση με την οποία μας, ε, μας βλέπουν. Κάποιοι που είναι πλούσιοι αλλά που Μα επιβάλλουν μια ιδέα ανάπτυξη που δεν, δεν, δεν μπορούν καν να μα την αναλύσουν, να μα πούν την αλήθεια. Άρα, η κρίση είναι μια ευκαιρία, ούτω ώστε να άρουμε όλη αυτή την κατάσταση, αυτή την ιονία ανάπτυξη που δεν μα επιτρέπει να κάνουμε κάτι από όλε μα τι πρώτε ύλε, να έχουμε την προσθέμενη αξία, αυτή την ε, επιβαλλόμενη δημοκρατία που επιβλήθηκε από αλλού και να λέμε να εμεί ψηφίζουμε για άλλου. και έτσι να νομιμοποιούμε μια ηγετική τάξη που μετά συνεχίζει στον ίδιο δρόμο του νεοφιλελευθερισμού που καταστρέφει απασχόληση, γεωργία και αυτή την όποια βιομηχανία έχουμε. Τις παραδοσιακές τέχνες, όλα, τον πολιτισμό και εγώ σαν γυναίκα αισθάνομαι απελπισία γιατί οι γυναίκες παίρνουν με τη ζωή τους αυτή την κατάσταση. Και η Αφρική στέκεται στα πόδια της γιατί οι γυναίκες είναι στο πόδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στις επάλξεις. Τι γίνεται με την Παγκόσμια Τράπεζα. Με κάθε σεβασμό. Αγαπητέ. Δεν είναι προσωπικό το θέμα κύριε Πλάντο όμως αυτό είναι ένα ερώτημα που όλοι θα πρέπει να το θέσουν. Τι θα αποτύχουμε κι εμείς όπως θα πέτυχαν όλοι οι άλλοι ή πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το σύστημα το οποίο δεν τα καταφέρνει. Υπότιτλοι ότι είναι μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη και που μας δημιουργεί πρόβλημα το οποίο έχει αποκτήσει τις διαστάσεις της παγκόσμιας. Κοιτάξτε λοιπόν τι έχουν πάθει οι Αφρικανοί. Θα πρέπει να αλλάξουμε επομένως κριτήρια το Δινέζο Νομικό Ταμείο να σταματήσει να ορίζει τις τύχες της Επίρου μας. Γιατί βλέπουμε ότι αποφασίζει το Δινέζο Μισματικό Ταμείο αντί για τους Αφρικανούς, για τους Αφρικανούς και τις Αφρικανές. Όμως το θέμα δεν είναι τι κάνει το Ταμείο, αλλά τι κάνει και η Ευρώπη, η φιλελεύθερη Ευρώπη που σήμερα γιορτάζει την πτώση του, του τείχους του Βερολίνου, μια που ορθώνονται άλλα τείχη. Είμαστε περικυκλωμένοι από τείχη. Για να ρωτήσουμε το G20 και το ΑΕΠ και οι δείκτες οικονομικοί και αυτό δεν είναι τείχος. Έτσι είναι ένας τείχος που δεν μας αφήνει να μπούμε στο κλαμπ των ισχυρών. Χρειάζεται επομένω στον ΟΗΕ κάτι σαν πραξικόπημα. Κάποιο εκεί να κάτσει και να του πει. Τι δεν έχει καλό. Το θέμα είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση. Πότε δεν υπήρχε σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό, ούτε θα υπάρξει δημοκρατία. Εάν δεν φροντίσουμε για κάποιες σωστές σχέσεις μεταξύ πλουσίων χωρών, αναγκαμένων χωρών, ε, των, των θεσμικών οργάνων και όλων των υπολείπων. Και σας το λέω αυτό γιατί για μια χώρα που έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι, είναι παγιδευμένη, το, το μισό είναι μια έρημος και τα παιδιά δεν έχουμε τι να κάνουμε, τι να ζήσουμε, και πρέπει να φύγουν. Νομίζω ότι έχει γίνει ο κόσμος μια τεράστια φυλακή. έχουν κλειστεί σε φυλακή πλούσια και έχουμε αυτές τις συμφωνίες της επανεισδοχής και έτσι είναι σαν δεσμοφύλακες οι ηγέτες των χωρών αυτών όσον αφορά τους μετανάστες. Και δεν διαδόψουν αυτό είναι ένα έγκλημα. και οι ερετοί μας άρχοντες ωφελούνται από αυτό. Το δε τίμημα το πληρώνουν οι Αφρικανοί και πιο συγκεκριμένα οι Αφρικανές. Ευχαριστώ. Muchas ευχαριστώ πολύ κυρία Τραωρέ. Και τώρα οι ευρωβουλευτές μπορούν να τοποθετηθούν ή να θέσουν ερωτήσεις εις τους ε, εμπειρογνώμονες, τους τόσο εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα. Έχετε το λόγο. Κάποιο Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει. Δεν ήμουν έτοιμος μετά τα πυροτεχνήματα της κυρίας Τραωρέ βέβαια έμεινα άναυδος ακούγοντας αυτές τις διαπιστώσεις και τις κατηγορίες που εξτόμισε. Ήθελα λοιπόν να θέσω ερωτήματα και στους δύο συμμετέχοντες. Για τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και παρά την αντίφαση που είδαμε για την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πρώτων συμμετεχόντων, ήθελα να μου πείτε Ερώτημα είναι. Κατά πόσο συμμερίζεστε τις δηλώσεις της κυρίας Αμενάτα Τραωρέ. Μεταξύ του όλου και του δίποτα υπάρχουν ε, δυνατότητες να δράσει κανείς. Εγώ είμαι μέρος της τάσης της μεταρρυθμιστικής. Θα μπορούσε κανείς να βελτιώσει τα πράγματα βάσει των εφιστάμενων υποδομών. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει ολοσχερός να καταδικάσουμε το FMI. Ξέρω ότι οι πολιτικές των, της δεκαετίας του 80 είχαν τις επιπτώσεις που αναφέρατε στην Αφρική, άλλωστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άλλαξε κάποια στιγμή η πολιτική, κατηγορήθηκε για τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και δημοσιονομικής ισορροπίας, τα οποία αυτά καθεαυτά δεν ήταν αρνητικά, διότι η δημοσιονομική ισορροπία δεν ήταν κάτι αρνητικό, αλλά αυτό που πάντοτε μας απασχολούσε και υποδεικνύαμε ήταν η έλλειψη παρακολούθησης των πολιτικών του FMI. E. Εάν δεν υπάρξει πολιτική μεταρρύθμιση δεν υπάρχει και υλοποίηση των πολιτικών του ΕΦΜΗ. Αν δεν υπάρξουν κοινωνικέ αλλαγέ, το ΕΦΜΗ θα διδραματίσει το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Και εδώ και ω προ του δανειστέ ε, υπάρχει ένα θέμα οι οποίοι είχαν από τη δεκαετία του 70 δεσμευτεί να, ε, να εκταμιεύσουν 0,7 του ΑΕΠ Το 2005 αναλήφθησαν νέες υποχρεώσει και σήμερα μας ρωτάνε τι έγινε με αυτές τις υποχρεώσει που αναλάβατε το 2005. Φαίνεται ότι οι υποσχέσει αυτές δεν θα κρατηθούν. Και μια άλλη ερώτηση προς την κυρία Τραωρέ. Τα υπάρχοντα κείμενα από τις συμφωνίες του Σκοτονού που θα αναθεωρηθούν δεν περιέχουν βάσεις τέτοιες που να επιτρέψουν να χαράξουμε μια άλλη πολιτική. Η Συμφωνία της Κοτονού προβλέπει την δράση νέων φορέων, όπως του ιδιωτικού τομέα ή της κοινωνίας των πολιτών ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Αφρική. Και ξέρουμε πώς έχει αντιταχθεί η Αφρική στην ε, συμπερίληψη της αναφοράς αυτής της κοινωνία των πολιτών στις συμφωνίες ε, της Κοτονού. Εάν λοιπόν σωστά κατάλαβα το νόημα τη ομιλία σα, σωστά έχει επιμείνει τότε για την συμπεριλήψη τη κοινωνία των πολιτών η Ευρώπη. Διότι η κοινωνία των πολιτών στην Αφρική θα πρέπει να προβλέψει τι δομέ τη χώρα που δεν έχουν αρκετή διακυβέρνηση. Διότι χωρί διακυβέρνηση το κράτο δεν μπορεί να αντιποκριθεί στι βασικέ αρμοδιότητε. Δηλαδή την διασφάλιση των πολιτών, την ασφάλεια του κράτου και τη κοινωνία και η Ένδια έχει πάρει το πάνω χέρι σε αυτές τις χώρες. Η Ένδια κυβερνάει, όπως το είπατε κι εσείς. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Προσπαθώ να βρω κομμάτια για να, τις ψηφίδες για να, κατα... για να συνθέσω αυτό το μεγάλο ψηφιδωτό, το πανόραμα του... που μας παρουσιάσατε στην ομιλία σας. Διότι εμεί ω πολιτικοί ηθήνοντε δεν μπορούμε να παραμένουμε χωρί απάντηση μετά από τόσα ζωφερά που μας περιγράψατε. Euh, Κυρία Τραωρέ, να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να βοηθήσει την Αφρική. Την τελευταία φορά όμως που κοίταξα τους αριθμούς, στα μέσα του Σεπτέμβρη, Είχαμε 1,60% των δανείων που προβλέθησαν προς όφελος της Αφρικής. Ήθελα λοιπόν να γνωρίζω επακριβώς τον κατάλογο των χωρών και τα ποσά τα οποία από τον μήνα Απρίλιο ωφελήθηκαν από τα κονδύλια του FMI. Τα 250 δις δολάρια και τα 750 δις δολάρια. Ποιο ήταν το μερίδιο που πραγματικά πήγε στην Αφρική. Ο κύριος Κάσμαρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υπερασπιστώ τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με όσα υπόθηκαν. Η δημοκρατία δεν μπορεί να αποδυναμώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Εάν βέβαια μιλήσει καλής, κανείς για τη Γερμανία, ο εκδημοκρατισμός δεν ευνόησε την οικονομική ανάπτυξη, δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Γιορτάζοντας τώρα τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, πρέπει να θυμόμαστε ότι 1,5 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι μετακινήθηκαν από την Ανατολική Γερμανία στην τότε Δυτική και ο μέσος μισθό παραμένει χαμηλότερο στα ανατολικά παρά στα δυτικά της Γερμανίας. Οπότε ο εκδημοκρατισμό δεν είναι πανάκια. Δεν είναι λύση για κάθε πρόβλημα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που ήταν φτωχή. Μια χώρα όπου οι μεταρρυθμίσεις, οι οικονομικές αλλαγές οφείλονται στην εισαγωγή της δημοκρατίας, αλλά δεν είναι πανάκια η δημοκρατία. Είναι μια επιπλέον βοήθεια, αλλά δεν είναι λύση σε κάθε πρόβλημα. Όταν μιλάμε για το άχθος, τις δημοκρατικές δυνατότητες, τους τοπικούς πολιτικούς ηγέτες, αυτοί θα έπρεπε να διαθέτουν εργαλεία ώστε το δημοκρατικό δυναμικό να αξιοποιείται. Νομίζω όμως ότι μια παράβατη εδώ συνθήκη είναι η συμμετοχή των ίδιων των λαών, των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή δημοκρατική νομιμότητα δεν έχουν καταφέρει παρόλα αυτά να λύσουν τα οικονομικά προβλήματα των χωρών τους. Βεβαίως μπορούμε να λέμε ότι είμαστε υπερβολικά αργοί. Γι' αυτό δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου η ευθύνη της δημοκρατίας. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που έφτασα στο τέλος της ομιλίας της κυρίας Τραωρέ. Έχασα τις ομιλίες σχεδόν ολόκληρες. Αλλά έχοντας, αφού σας άκουσα νομίζω ότι μπορώ να παρέμβω και σας ευχαριστώ που μας μιλήσατε με τρόπο τόσο ειλικρινή και ευθύ στις... και ζωφερό. Σε αυτό το σώμα έρχονται πολλοί και μας μιλούν ε, για να ακούσουμε αυτά που μας αρέσουν, θεωρούν με γλώσσα διπλωματική και αυτή τέτοια που να χαϊδεύει τα αισθήματά μας και να μπορούμε να καταπιούμε εύκολα τα λεγόμενά τους. Πολλοί μιλούν εδώ για δημοκρατία στο Κοινοβούλιο. Αλλά τι προσφέρει η δημοκρατία αν δεν γεμίζει τα στομάχια, εάν δεν δίνει νερό σε ένα παιδί, ε, φάρμακα στα παιδιά ή σε μια γυναίκα που μπορεί να πεθάνει στη γέννα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί και η ίδια η δημοκρατία μετά τις αλλαγές για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών προσφέρουν πραγματικά την αξιοπρέπεια. Έχετε δίκιο. Ε, γύρουμε φραγμούς κεφαλαιοχικούς, επενδυτικούς, ενθαρρύνουμε τις επιχορηγήσεις, όταν έχουμε υπερπαραγωγή κάποιου προϊόντος, μετά πηγαίνουμε στις αναπτυσσόμενες αγορές, ε, χώρες και οδηγούμε σε πτώχευση τις αγορές τους. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να δούμε τους εαυτούς μας πριν κατηγορήσουμε τους υπόλοιπους. Για τη μετανάστευση όλοι ε, στο κοινοβούλιο φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται ακριβώ τι σημαίνει μετανάστευση. Πάντοτε θα υπάρχει μετανάστευση εφόσον κάποιοι δεν δέχονται να μην διεκδικήσουν μια καλύτερη διαβίωση για τον εαυτό τους ή για αυτούς που αφήνουν πίσω τους. Μην ξεχνάμε ότι τα εμβάσματα αποστέλλονται στις αναπτυσσόμενες χώρες μακριά πέρα από τις θάλασσες και ανεξάρτητα από την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα σταματήσουμε λοιπόν αυτές οι μεταναστευτικές ροές μόνο να αντιμετωπίσουμε τα μείζωνα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Τις επενδύσεις, τις τραγικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που δεν βρίσκονται στο μακρινό μέλλον, αλλά ήδη λαμβάνουν χώρα. Και όταν αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να εξαλείψουμε τη φτώχεια, τα βασανιστήρια, τους πολέμους και την, ε, και την κακή διαβίωση. Αυτό είναι κάτι που οδηγεί επίσης τους ανθρώπους να διαφεύγουν από τις χώρες τους. Παρακαλούμε συνεχίστε να μας μιλάτε σε αυτόν τον τρόπο, συνεχίστε να δράτε όπως κάνατε. Μην ωρεοποιήσετε και μην εξοραίζετε καθόλου τα λόγια σας και τι ομιλίε σας. Διότι μην ξεχνάτε ότι κάποιες φορές υπήρχε τη Βαβέλ καταραίων τελικά. Για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να πω ότι ήμασταν εδώ όταν είχαμε μια εξαιρετική έκθεση που είχε ετοιμάσει για μα ο καθηγητή Νάιρι Woods, η οποία κάλυπτε το θέμα των εμβασμάτων και τα νέα κονδύλια που διατίθενταν ε, λόγω της οικονομικής, της οικονομικής κρίσης. Μια κρίση που προκάλεσε η απληστία κάποιων και την οποία βέβαια υπέστησαν, υπέστησαν αυτοί που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, αυτοί που ήταν οι πλέον αδύναμοι. Πρόεδρε, είναι ενοχλητικά χαμηλό το ποσοστό των κονδυλίων που δανείστηκαν στην Αφρική σε αυτή την περίοδο. 86% ε, ε, των κονδυλίων αυτών κατευθύνθηκαν στις λεγόμενες αναδυόμενες δημοκρατίες. Ε, πέρα από λοιπόν από αυτήν την απάντηση, θα ήθελα μια απάντηση για το αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα μήπως ήταν καλύτεροι στο έργο τους αν είχαν μια ευρύτερη αντιπροσωπευτική βάση. Και εμεί ω βουλευτέ, τι θα πρέπει να ζητήσουμε ώστε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να μπορεί να αντιμετωπίσει τα επικριτικά σχόλια που τόσο συχνά το απευθύνονται. Πάντω, αυτό που σα είπα δεν το εννοούσα ω φιλοφρόνηση, κυρία Τραωρέ. Το θεωρώ δεδομένο. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δεν φαντάζονται. Τι είναι να βλέπει κανείς το παιδί του, το μοναχογιό του, να εγκαταλείπει τη χώρα του για το μόνο και απλό λόγο ότι το μέλλον του είναι αβέβαιο. Μπορεί να πεθάνει, να ζει σε συνθήκες πείνας που ούτως ή άλλως θα τον οδηγήσουν στο θάνατο και νομίζω από την άποψη μιας μητέρας ή μιας γυναίκας αυτό καλό είναι να αντυχήσει εδώ στους τοίχους του Ευρωκοινοβουλίου και να φτάσει και στα αυτιά των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Αν δεν έχουμε άλλε ερωτήσει, θα ήθελα και εγώ ίδιο να υποβάλω μία. Ε, στις ε, δύο αυτές ε, εισηγήσεις ακούσαμε κάτι για το Διανέργο μερικό Ταμείο πριν από μία πενταετία θα θεωρεί αδιανόητο. Μας είπαν ότι είναι τόσο μεγάλη κρίση που θα πρέπει να δείξουμε κάποια ελαστικότητα όσον αφορά τους νομισματικούς αλλά και δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό είναι καταρχήν ε, παράδοξο, αυτό είναι καταρχήν ερετικό σε σχέση με την ιστορία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε σχέση με το χαρακτήρα της κρίσης η οποία σοβεί και στη συνέχεια η κυρία Τραωρέ, Μας είπε η κυρία Τραωρέ ότι ορισμένα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά χτυπητά τα οποία θέλω να σας τα επισημάνω ότι είναι πάγια, συνεχής η κρίση, ότι δεν ε, ήρθε τώρα, δεν είναι συνέχεια της κρίσης του 2008, αλλά ότι είναι συνεχής και μας επισήμανε ότι κάποια βήματα πρόοδου τα οποία σημειώθηκαν στο παρελθόν και τα οποία ίσως θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πεδίο της μακροοικονομίας δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τη ζωή του Κοσμάκη και επίσης ανέφερε και κάτι άλλο ακόμα πιο έντονο, πιο, πιο εντυπωσιακό ότι αυτοί γίνονται μάρτυρες, μάρτυρες που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μιας νέας κατάτμισης διαμελισμού της Αφρικής και συμπερίστε, συμπαθάτε με γι' αυτό αλλά νιώθω κι εγώ τόσο μεγάλη γανακτήση που τελικά από, μέσα από εκεί βρίσκουμε την ενέργεια για μια αλλαγή οπότε μπορεί να ξεκινήσει κάτι αν αρχίσουμε να παλεύουμε στη συνέπεια αυτής της βαθιάς κρίσης που τόσο πολύ έχει πλήξει τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Los ponentes tienen cinco minutos eh, cada uno. Οι συμπτές μας έχουν ένα πεντάλεπτο έκαστος, ούτως ώστε να σχολιάσουν τις ερωτήσεις. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε, ήθελα να ξεκινήσω με μια αστεία ιστορία, κάτι που σκέφτηκα και πριν από την κρίση την ίδια. Μιλούσα με έναν πρόεδρο Αφρικανικής χώρας, ο οποίος θεωρούσε ότι τα κονδύλια του έχουν ε, πάρει λάθος δρόμο, δεν ήξερε που πήγαιναν, ποιο τα έπαιρνε και αυτό ισχύει για πολλές χώρες που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις με λιγοστούς τους πόρους. Ε, του εξήγησα τη μακρονομική άποψη ως προς αυτά. Ε, κατάλαβε, ήταν έξυπνο και έγνεψε, αλλά μου γύρισε και μου είπε ωραία είναι όλα αυτά τα μακροοικονομικά. Αλλά έχετε τίποτα τρακτέρ για μας. Έμεινα κάπως άναυδος και του είπα είμαστε από το Διεθνές Μαρματικό Ταμείο. Όχι, μου είπε. Δεν θέλω άλλα χρήματα. Ο Υπουργό Οικονομικών μου θα τα κλέψει αν μου τα δώσετε. Δώστε μου κάτι που πραγματικά να έχω ανάγκη. Τρακτέρ. Νομίζω ότι αυτό το περιστατικό Μα δείχνει τρει ιδέε. Πρώτα απ' όλα ότι η ανάπτυξη χρειάζεται μακροοικονομική σταθερότητα. Πρέπει επίση οι δημοσιονομικοί περιορισμοί να αντιμετωπιστούν από του υπευθύνου και να γίνουν και επιλογέ οι χώρες που δεν περνούν σε αυτή τη διαδικασία θα αφήσουν άλλους να αποφασίζουν εκ μέρους τους και αυτό δεν μπορεί να το επιτρέψει κανείς. Χρειάζεται λοιπόν να έχει κανεί και τα τρακτέρ αλλά και τη μακροοικονομική πολιτική που θα επιτρέψει να υλοποιήσει την αναπτυξιακή βοήθεια, να τη χρησιμοποιήσει. Δεν ήθελε άλλα χρήματα ο άνθρωπο, ήθελε κάτι πραγματικό. Και ο ίδιο υπέδειξε του υπευθύνου τη διαφθορά. Το να δίνει κανεί χρήματα σε ένα σύστημα διεφθαρμένο δεν πρόκειται να παράγει τρακτέρ. Αλλά τέτοιου είδους μαθήματα είναι αυτά που πρέπει να μάθουμε. Το, η διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα έχει μάθει με δυσκολία ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που μας είπε η κυρία Τραωρέ για τη δεκαετία του 80 και 90 είναι σημαντικά. Μπορεί να ακολουθήσαμε τον δρόμο της αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά δεν μειώσαμε τη φτώχεια, δεν καταπολεμήσαμε την ε, έλλειψη δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν ε, να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που δρούμε από τη δεκαετία του και το κάναμε αυτό. Επικεντρωθήκαμε σε δύο συγκεκριμένα χώρε που μα λένε πώ αυτέ θέλουν να αναπτυχθούν. Μα είπαν ποιε είναι οι στρατηγικέ του καταπολεμήσει τη φτώχεια και εμεί αποφασίσαμε να τι χρηματοδοτήσουμε. Και μάλιστα ανακουφίζοντά τι από το χρέο και θέτοντα στόχου αναπτυξιακού. Έτσι αρχίσαμε να κατασκευάσουμε μια αμερόληπτη και ίσω αδιάφθορη στρατηγική ανάπτυξη για τον κόσμο. Όμω όταν αρχίσαμε να ακούμε τις φωνές ε, των ανθρώπων όπως η κυρία Τραωρέ, αποφασίσαμε ότι πρέπει να ακούγονται και αυτές οι φωνές. Μπορεί να μην έχουμε τις απαντήσεις, αλλά στη διεθνή κοινότητα κάναμε κάποια πρώτα βήματα για να ακούσουμε τους ανθρώπους, να ακούσουμε τις ανάγκες της τοπικής ανάπτυξης, τις τοπικές φωνές που θέλουν να στηρίξουν την ε, ανάπτυξη. Αυτέ είναι οι πρόσφατε εξελίξει. Είναι αργέ. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να πάμε και πιο γρήγορα. σω θα έπρεπε να έχουμε όλε τι απαντήσει, αλλά υπάρχει μια καθοριστική στροφή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την αναπτυξιακή βοήθεια και την ε, δράση μας. Από τη μακρονομική προοπτική να δούμε μόνο είναι περιττό. Σήμερα έχουμε αλλάξει άποψη για το ποιο είναι ο σωστό τρόπο να αναπτυσσόμαστε, ποιοι είναι οι σωστοί μηχανισμοί. Δεν υπήρξε καμία χώρα παγκοσμίω που να μην καταπολέμησε σημαντικά τη φτώχεια χωρί τη μέτρηση τη ανάπτυξη λόγου χάρη. Η ανάπτυξη χρειάζεται, αλλά δεν είναι αρκετή. Δεν αρκεί για να ταΐσει κανείς τους ανθρώπους, για να τους προσφέρει εκπαίδευση, για να τους δώσει υγειονομικές υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρξει αύξηση μακροοικονομική ε, σταθερότητα στους αριθμούς. Χρειάζονται και οι θεσμοί που θα υλοποιήσουν τις στρατηγικές. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε τους λαούς. Και ε, νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει πρόοδο στην πράξη και θα συνεχίσουμε. Όσο περισσότεροι άνθρωποι σαν την κυρία Τραωρέ ε, μιλούν, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρνουμε. Επίσης, μια ερώτηση του Πρόεδρου και ενό άλλου μέλους για το ποσό τη βοηθειά μα. Δεν έχω του ακριβεί αριθμού μπροστά μου, κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να του φέρω αν του χρειάζεται η Επιτροπή σα, αλλά μιλάμε για ποσοστό για το κονδύλια που στέλνουμε στην Αφρική χαμηλό σε σχέση με το τι εκταμιεύει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για άλλε χώρε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η φύση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου του ίδιου είναι ιδιαίτερη. Σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα συλλογισμού που είναι οξύτατα και έχουν συστημικές επιπτώσει για τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε αναπτυξιακό οργανισμό που εργάζεται στην Αφρική μόνον και εφόσον οι χώρε που βοηθούμε ασχολούνται με μακροοικονομικές ελλείψει ισορροπία. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Για να έχουμε ανάπτυξη στην Αφρική χρειάζεται χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις. Πρέπει κανείς να επενδύσει καιρό στο ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν αρκεί για να τα καταφέρει αυτά. Διότι και εμείς χρηματοδοτούμαστε από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλους δωρητές με πολύ ισχυρή φωνή έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε κάποιες ελάχιστες δεσμεύσεις ε, και να τις αναλάβουν οι υπεύθυνοί μας. Ε, εάν δώσει ένα ποσοστό η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και του τάξη το 0,7% κάτι θα καταφέρουμε. Όμως μπορείτε να πείτε ότι σε κάποιες χώρες απλά μπαλώνουμε ε, τα κενά αλλά είδαμε σε άλλε χώρε να αναπτύσσονται πραγματικέ αναπτυξιακέ στρατηγικέ. Οι πόροι ήταν περιορισμένοι. Οι χώρε βασίστηκαν στο δεδομένο ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι χαμηλή ότι τα ποσά που υποσχέθηκε το G7 και η διεθνή κοινότητα γενικότερα τελικά κατέληξαν να είναι πολύ χαμηλότερα. Και θα πρέπει να βάζουμε επιδέσμου και να πουλώνουμε τέτοιε πληγέ εφόσον τα προβλήματα συνεχίζουν να τρέχουν, εφόσον ο κόσμο δεν αποφασίζει να στηρίξει την ανάπτυξη. Σωστή είναι η έκκληση, η έκκληση για περισσότερα χρήματα για την Αφρική, για περισσότερη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ποια θεσμικά όργανα είναι αυτά που πρέπει να δώσουν τα κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τι αφρικανικέ χώρε με τον σωστό τρόπο, άρα να πληρώσουμε και το κόστο. Δεν είναι όμω υπεύθυνο το θεσμικό όργανο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για αυτό το σκοπό. Και για τη δημοκρατική βάση, πρόεδρε, να κάνω ένα σχόλιο για την ε, αντιπροσώπευση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που απηχεί στα αυτιά του κόσμου. Το G20 συζήτησε γι' αυτό. Είναι πολλά όσα πρέπει να γίνουν για την κατανομή των ψήφων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζουμε ότι ως το 2011 θα έχουμε ολοκληρώσει τη μεταρρύθμισή μας και ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Κυρία Τραωρέα, για πέντε λεπτά. Donc, euh, Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας των όσων πιστεύουν ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Σε παγκόσμια κλίμακα και για πρώτη φορά και στο βορρά όπως και στο νότο όλοι πλησόμαστε από αυτή την δυσμένη συγκυρία. Κάτι το οποίο απορρέει από την συγκέντρωση των πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών μέσων για τον ΜΜΕ και από το από το ότι γίνεται αυτή η, συγκέντρωση χωρίς κανένα όριο. Και βεβαίως βεβαίως και ξέρω ότι υπάρχει ωραία που λέει ότι φταίει η φτώχεια, ναι, αλλά η φτώχεια δεν είναι και το νομοτελειακό. Η φτωχή είναι θύματα του πλούτου. και όλοι μαζί μέσω του δουλεμπορίου, στήριξαμε τον καπιταλισμό με την απεικιοκρατία και επομένω η έξοδος από την κρίση είναι κάτι το οποίο περνάμε μέσα από την Αφρική. Δεν, θέλω άλλο να, να λυπόμαστε τους Αμερικανούς και να λέμε ότι α, εκεί κάτι να κάνουμε για να, να, να, να, να βελτιώσουμε τους Αμερικανούς. Ας αλλάξουμε οπτική γωνία, να αλλάξουν νοοτροπία, σταματήσει αυτή η λύπηση. Εμείς οι ίδιοι με την διαφθορά, με την ανικανότητα της ηγετικής τάξης εδώ και τόσο καιρό, ε, χάσαμε το δικαίωμα του να κοιτάμε τους άλλους επίσης ώρες. 12 εκατομμύρια σου έχει η χώρα μου. 127 όμως κόμματα. 250 στο Κονγκό. Και εάν κανείς θέλει να είναι σοβαρός, θα πρέπει να δει πώς μπορεί να υπάρχει κάποιο δομημένη άποψη για τις σημερινέ προκλήσεις οικονομικές, οικολογικές, πολιτικές. Εδώ όμως δεν υπάρχει όραμα στην Αφρική και με αυτά, με αυτές τις αντίσεις βγαίνει κάτι. τελευταίες ε, δεκαετίες χαμένα σωρός αντίς κορυφής για ό,τι θέλετε. Κανένα όμω πια δεν πιστεύει ότι έτσι θα βρεθεί κάποια λύση. Κοινωνική συνέντευξη κορυφή, για τι γυναίκε κλπ. Ε, αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το μηδέν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και αυτή η στόχη, η αναπτυξιακή τη χιλιετία, που δεν υπάρχει καμία τύχη. Καμία πιθανότητα να τις πετύχουμε. Θα πρέπει να Γυρίσουμε σελίδα. Βάζω για το λιθαράκι μου. Με μια προσπάθεια για τη χώρα μου. Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξη. Δεν δικαιούμαι να είμαι απεσιόδοξη. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παιδαγωγικό με κάποια μικροπρογράμματα. Προσπαθώ να δημιουργήσω προβληματισμό για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για μας. Και όλα αυτά τα οποία σωρεύουμε ως εναλλικές λύσεις δεν ενδιαφέρουν κανένα. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρει την ε, άρχουσα τάξη είναι να διατηρήσει αυτή την ιδιότητά της, να ωφελείται. Είναι στο γόνατο αυτή η ανάπτυξη φτιαγμένη. Και η δημοκρατία μας επίσης στο γόνατο φτιάχτηκε. Το θέμα δεν είναι τι κάνει το νομισματικό ταμείο, είναι το να μπορέσουν οι ίδιοι Αφρικανοί να ξέρουν τι θέλουν, να σκεφτούν τι θέλουν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, όλα όσα κάνουμε μας, μας ε, διαιρούν. Έχουμε αυτές τις κυρώσεις, ξέρουμε πού προέρχονται, ξέρουμε τι κάνουν ή τις άργουσες τάξεις. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι η πιο σημαντική πρωτήλη. Οι άνθρωποι. Και κερδισμένοι βγαίνουν άλλοι. Άλλο η Ευρώπη που οχυρώνεται θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι πάντοτε βασιζόταν στην ε, Αφρική γιατί είπαν τις πρώτες αλλά ταυτόχρονα ήταν η Αφρική και το κράτος των αχρήστων. Τα παιδιά πάνε και ασχολούνται με τα παλιοσίδρα, με σκουπίδια και αυτό δεν το λέω για να βρίσουν να κατηγορήσω κάποιον, όμως διαπιστώνω ότι τις τελευταίες μέρες αν δούμε τι ε, τι λέγεται, τι αισθάνεται ο κόσμος στη Γερμανία, τότε εγώ σκέφτομαι ότι ήταν σύμβολο ο τείχος, έπεσε, όμως εγώ λέω ότι έπεσε μόνο από πλευρά πρακτικής, γιατί στην ουσία υπάρχει ακόμα ο τείχος, όπως ήταν πριν η Ανατολή Γερμανία, τώρα είναι η Αφρικανή. Επανενώθηκε η Γερμανία, οικοδομείται η Ευρώπη, Έχουμε την ελεύθερη Ευρώπη και τις δημοκρατίες όμως ουσιαστικά έπρεπε να δει ότι το πρόβλημα που είχε παλιά η Ευρώπη τώρα το μετέθεσε στην Αφρική και οι Αφρικάνοι τώρα χτυπάνε την πόρτα στην Ευρώπη. Αλλά που να λύσει το πρόβλημά μας αφού καλείτε τους ηγέτες μας και τους λέτε να πάνε σε περαιτέρω φιλελευθεροποίηση και απορρίθμιση. Περισσότερος προστατευτισμός με την Κοτονού. Προστατευτισμός όμως για ποιον. Χρειαζόταν προστατευτισμός για τους πιο ευάλωτους. Δεν λέω να δώσετε τις απαντήσεις, εμείς πρέπει να τις δώσουμε. Και βλέπω, εδώ να χύνεται το γάλα, βλέπω τις αυτοκτονίες στη Γαλλία και λέω υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα και δεν φταίει η ανικανότητα των Αφρικανών. Θα πρέπει σε όλο τον κόσμο να το εξετάσουν το πρόβλημα και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε τη διέξοδο. Ο πρόεδρο. Ευχαριστώ και του δύο συγκητέ οι οποίοι μα παρουσίασαν κάτι τόσο ενδιαφέρον. Επόμενος γύρος τραπέζι τώρα. Ξεκινά δεν ξέρω αν θα το προτείνω όπως πρέπει. Πρόκειται από την Νορβηγία. Σέλντερουπ. Μπορείτε να κάνετε την εισήγησή σας για 25-30 λεπτά. Uh, thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Uh... Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ μιλώ εκ μέρου τη ε, Νορβηγική Επιτροπή που ασχολήθηκε με τη φοροδιαφυγή και τι επιπτώσει τη ε, στην ανάπτυξη. Η εντολή που είχαμε από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο ήταν να καταμετρήσουμε τη διαφυγή των παράνομων κεφαλαίων και τις επιπτώσεις που, στην, που είχαν στην ανάπτυξη και να προβλέψουμε μέτρα για τις δυσμενείς επιπτώσεις που ενδεχομένως τα είχαμε εντοπίσει. Και τέλος να συντάξουμε συστάσεις που να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο της ανάπτυξης. Για τους φαρολογικούς παραδείσους και το πώς λειτουργούν. Επιτρέψτε μου να σας κάνω ένα σύντομο μάθημα να σας δώσω μια σύντομη διάλεξη για το θέμα αυτό, για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ε, επίσης τη σύμφωνη γνώμη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που έχουν διαβάσει την έκθεση και εγκρίνουν όλα όσα λέγονται. Κάποια αριθμή πρώτα απ' όλα η Επιτροπή μας διαπίστωσε ότι οι παράνομες κεφαλοκικές ροές εκτιμώντας τα 631.000 941 ε, δις αμερικανικά δολάρια. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι προς τις ε, φτωχότερες χώρες ε, αυτό το ποσό ξεπερνά την ε, εισρωή νόμιμων κεφαλαίων προς τις φτωχές χώρες και είναι 10 φορές μεγαλύτερο από την αναπτυξιακή βοήθεια που λαμβάνουν. Επίσης, αντιαπιστώσαμε ότι οι πλούσιότεροι μπορούν να κρύψουν τα κεφάλαιά τους σε φορολογικούς παραδείσους σε ποσό που ανέρχεται στο ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, 20% αυτών των κρυμμένων κεφαλαίων κρύβονται από τις άρχουσες τάξεις, τις ηθήνουσες τάξεις της ε, φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό από μακρονομικής άποψης σημαίνει ότι η κυβερνόσα τάξη στις φτωχότερες χώρες υπερεκπροσωπείται στο επίπεδο των φορολογικών παραδείσων. Επίσης, οι πλουσιότεροι των δυτικών χωρών δηλώνουν μόνο 5% αυτού που πραγματικά καταθέτουν στους ε, φορολογικούς παραδείσους. Και αυτό βεβαίως έχει και μια διάσταση αναδιανομής των κεφαλαίων, την οποία θα σχολιάσω σήμερα. Τώρα, γιατί ξεχωρίζουν οι φορολογικοί παράδεισοι από αυτά που έχουμε ονομάσει νόμιμα κράτη. Έχουμε Έχουμε μια σειρά από βιβλία για αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους και έχουμε τις υψηλές φορολογίες και τις κανονικές ρυθμίσεις. Έχουμε εταιρείε που ακολουθούν συγκεκριμένη συμπεριφορά στα κράτη τους και υπάρχει φορολόγηση χαλαρή ή λιγότερο αυστηρή και μυστικότητα. Ή κάποιες φορές υπάρχει και απόρριτο οι επενδύσεις για τους ξένους επενδυτές. Οι έννοιες αυτές έχουν σκοπό να αποσπάσουν εισόδημα από τους ξένους επενδυτές και από τους φορολογητές. Η νομοθεσία για τους ξένους επενδυτές είναι τόσο καταστρεπτική που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από τις ε, ντόπιε εταιρείε. Η νομοθεσία επικεντρώνεται στις φορολογικές βάσεις άλλων χωρών. Εάν δούμε τώρα αυτές οι δικαιοδοσίες πώς λειτουργούν και πώς μπορούμε να τις συγκρίνουμε με νόμιμα κράτη, πρέπει να ξέρουμε ότι στα νόμιμα κράτη υπάρχουν δημόσια ε, μητρώα, υπάρχουν ε, τις αφροφυλάκια που ελέγχουν τα βιβλία των εταιριών, υπάρχουν λογιστικά πρότυπα, υπάρχει ισορροπή νομοθεσία που συγκρατεί όλο τον κοινωνικό ιστό. Η φορολογική παράδειση δεν έχουν τίποτα από αυτά. Έχουν ρήτρε διαφυγή που σημαίνει ότι αν κάποιο πάει στο φορολογικό παράδεισο και θελήσει να διερευνήσει κάτι, μπορεί τα κονδύλια αυτά να έχουν ήδη μετακινηθεί σε έναν επόμενο φορολογικό παράδεισο. Και συνεχώ υπάρχουν εξαιρέσει και ρήτρε διαφυγή. Η Επιτροπή μα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα παρατήρησε όλα αυτά και είναι ιδιαίτερα ε, επιφυλακτική για το κατά πόσο το G20 μπορεί να, λύσει, μπορεί να λύσει τα προβλήματα των ε, φορολογικών παραδείσων. Γιατί ακόμη και οι δομέ που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν ε, και η επαναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματο μαζί με την έλλειψη ενημέρωση και την απουσία μετρών σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία μαζί δεν πρόκειται να εξαλείψουν του φορολογικού παραδείσου μέσω των συνθήκων ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι ο Μπάρακ Ομπάμα στη φωτογραφία. κατά την προεκλογική του εκστρατεία και βρίσκεται έξω από το μεγαλύτερο, αυτό είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο για στοιχήματα και τζόγο. Είναι ένα μικρό κτίριο στο νησιά Κέιμαν όπου όμως 12,5 περίπου χιλιάδες εταιρείες έχουν την έδρα τους και οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους. Εδώ υπάρχουν κυρίως ταχυδρομικές θηρίδες και τα έσοδα που φτάνουν σε αυτό το σημείο έρχονται από άλλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι. Είναι εντυπωσιακό ότι το κέρδος αυτό δεν παράγεται στους νήσους Κέιμαν και ότι τα εισοδήματα αυτά που παράγονται αλλού δεν υπόκειται σε καμία φορολόγηση στους νήσους Κέιμαν, τώρα στις Βρετανικές Παρθένους νήσους. 19.000 κάτι και 830 καταχωρημένες εταιρείες με 43... 830.000 καταχωρημένες εταιρείες με 43 εταιρείες ανακεφαλή. Άλλη μια παρατήρηση. Η φορολογική παράδειση είναι πολύ μικρές δικαιοδοσίες με ελάχιστη με ελάχιστους διοκτήτες που ζουν αλλού, οι οποίοι δεν φορολογούν το κεφάλαιο και αν το φορολογούσαν, ακόμα και τις αναλλαγές να φορολογούσαν δεν θα είχαν κέρδος. Μιλούμε λοιπόν εδώ για το αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κλέφτη στην διαδικασία της φοροδιαφυγής και η απάντηση που θα σα έδιναν οι υπεύθυνοι του φορολογικού παραδείσου είναι ότι δεν θα απέδιδε κανένα κέρδο κάτω τέτοιο. Τώρα για τα σημαντικότερα συμπεράσματα τη Επιτροπή μα. Το πέμπτο και το έκτο συγκεκριμένα, η φορολογική παράδειση κάνουν τι εγκληματικέ δραστηριότητε πιο απλέ, διότι έχει κανεί ένα πιο ασφαλέ μέρο όπου μπορεί να κρύψει τα λάθηρά του. Εάν κάποιο καταφέρει ουσιαστικά να καλύψει έναν εγκληματία, είναι σαν να γίνεται συνεργό. Και το έκτο συμπέρασμα, μια ελκυστική πρόταση για όλου. Η μείωση των ε, φορολογικών υποχρεώσεων. Στον ε, τομέα των επίσημων ε, δραστηριοτήτων, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Επιτρέψτε μου να περάσω στα επόμενα σημεία. Η Νορβηγική Επιτροπή θεωρεί ότι οι φορολογικοί παράδεισοι πλήττουν την ε, ισορροπία των υπόλοιπων κρατών. Και γιατί το λέμε αυτό, Γιατί θεωρούμε ότι στο διεθνέ φορολογικό δίκαιο το εισόδημα θεωρείται ότι πρέπει να φορολογείται στη χώρα που παράγεται, όπου, από όπου προέρχεται. Αυτό είναι μια βασική έννοια. Και ότι οι ιδιοκτήτε πρέπει να φορολογούνται εκεί που εδρεύουν. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με αυτέ τι ταχυδρομικέ θηρίδε στα φορολογικού παραδείσου. Η Νορβηγική Επιτροπή λοιπόν ουσιαστικά λέει ότι η φορολογική παράδειση παρέχουν έδρα σε εταιρείε που λειτουργούν και δρούν σε άλλα κράτη και τις διαχειρίζονται άτομα που ζουν σε άλλα κράτη. Επίσης, αποκρύπτουν όλες τις πληροφορίες για, τους, ε, για τα μέλη των εταιριών και τους ιδιοκτήτες τους. Γιατί το κάνουν όμως αυτό. Είναι ελκυστική ακριβώς γιατί έχουν τέτοια νομοθεσία. Είναι ελκυστική η παράδειση αυτή για τους επενδυτές γιατί και έχουν ανάγκη και από συγκεκριμένα κεφάλαια. Και υπογράφουν φορολογικές, ε, οι επενδυτές υπογράφουν φορολογικές συνθήκε με τις φτωχότερες χώρες, οι οποίες δέχονται τέτοιες συνθήκες σε αντάλλαγμα κεφαλαίων. Εδώ να σας θυμίσω ότι ένας αρρώστος των συνθήκων αυτών είναι ότι το φόρος τελικά δεν πληρώνεται πουθενά. Στην Ινδία 57% των ξένων επενδύσεων προέρχονται από χώρες με πάρα πολύ μικρό πληθυσμό και πολύ μεγάλο κέρδος, πολλά μεγάλα κέρδη από την Νορβηγία. Πώς γίνεται αυτό. Αυτοί που ωφελούνται από αυτή την ισορροπία κεφαλαίων στην Ινδία είναι επενδυτέ και φορολογική παράδοση. Ε, Επίση, οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ πλύνονται από, τις του φορολογικού παραδείσου. Μα έδειξε η πρόσφατη κρίση ότι οι ε, φορολογική παράδεισοι ουσιαστικά εμποδίζουν του επενδυτέ να λειτουργήσουν κανονικά και νόμιμα, όπως οι επενδυτές μπορούν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και πληροφορίες. Τι σημαίνει αυτό για τις στοχότερες χώρες, ότι δεν, τα δάνεια για τις φτωχότερε χώρες γίνονται πιο ακριβά. Αυτός είναι ένας γνωστός μηχανισμός, τον οποίο έχουν σχολιάσει επανειλημμένως οι οικονομολόγοι. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η φορολογική παράδειση αυξήνουν και το κόστος τη φορολογία. Πώς γίνεται αυτό, όταν κανείς δεν μπορεί να φορολογήσει το κεφάλαιο, και αυτό γίνεται με τρόπο άδικο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στι αναπτυσσόμενε χώρε το φορολογικό κεφάλαιο είναι η σημαντικότερη πηγή εισοδήματο. Στην Ευρώπη, με την βιομηχανική επανάσταση, έχει αναφερθεί ότι σε χώρε με πληθυσμό κατώτερο των 20 εκατομμυρίων κατοίκων, τελικά το κεφάλαιο μπορεί να προέρχεται από 236 εταιρείε. Τι κάνουν λοιπόν οι χώρε αυτέ για να αντιμετωπίσουν τη μείωση από το φορολογικό κεφάλαιο που δεν λαμβάνουν. Επιβάλλουν υψηλότερου φόρου στην εναπομείνασα φορολογική βάση που διαθέτουν. Έτσι υπάρχει περισσότερο λαθρεμπόριο στις χώρες αυτές με τις εισαγωγές και εξαγωγές και όλα αυτά βεβαίως ε, παρεμποδίζουν και την ανάπτυξη. Επίσης η κατανομή των πόρων ε, δυσχεραίνεται, διότι οι φορολογικοί παράδεισοι κάνουν πιο ελκυστική τη μετακίνηση των ε, επενδύσεων σε τομείς που μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ωφελήματα των ε, φορολογικών παραδείσων. Μεγάλες εταιρείες κόβουν τους δεσμούς με τους φορολογητές και το κέρδος τους, φροντίζοντας να έχουν ε, ιδιαίτερα κερδοφόρα προγράμματα και αποδυναμώνοντας την αναδιανομή των ε, πόρων στις φτωχότερες χώρες. Τώρα να σας μιλήσω για μακρονομικά και δημοκρατία και θα σας παραπέμψω και στους δύο προηγούμενους ομιλητές. Μια από τις βασικές συνεισφορές ε, της ερευνητική αυτής επιτροπής είναι ότι η θεσμική σταθερότητα είναι σημαντικότερη για την οικονομική ανάπτυξη. Όταν μιλάω για θεσμική σταθερότητα, ενώ την καταπολέμηση της λαθοκρατίας, το κράτος δικαίου, τον εκδημοκρατισμό. Ξέρετε ότι για να βελτιωθεί η θεσμική ποιότητα και εφόσον διπλασιαστεί, διπλασιαστεί η θεσμική ποιότητα, μπορούμε να εφταπλασιάσουμε το εθνικό εισόδημα. Η Επιτροπή μας κατέληξε ότι η φορολογική παράδειση ε, κάνουν πιο ελκυστική και την ε, κλοπή πόρων από την κοινωνία, καθότι το λάθυρα μπορεί κανείς να τα κρύψει. Ασφαλώς αποδυναμένεται η θεσμική ποιότητα των φτωχότερων χωρών και δεν μπορεί να βελτιωθεί ο κοινωνικό του ιστό. Αυτό είναι βέβαια πολύ προβληματική τάση και το θέμα είναι αν μπορούμε να την ε, αντιμετωπίσουμε. Το να κλέβει κανεί τα χρήματα των φορολογουμένων σημαίνει λιγότερε επενδύσει στην ε, θεσμική ποιότητα. Ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό στο 1979 ένας από τους πιο πρόσφατους δικτάτορες τη δεκαετία του 70 έκλεψε περίπου 50 έως 80% του εθνικού προπολογισμού χρήματα τα οποία κρύφτηκαν σε φορολογικούς παραδείσους. Ως συνέπεια, το 92, ε, το κεφάλαιο της χώρας ήταν το μισό από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν η ανάπτυξη. Άλλα παραδείγματα. Ο Σερεμπακτα πρώην πρόεδρος. Υπεξίασε περίπου 3 δις δολάρια. Ο κύριος 10%, ο κύριος Ζαρντάρη. Σύζυγος της Μπούτου, πρόεδρος της ε, Πακιστάνου, ο κύριος 100%. 500 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Τουλάχιστον. Και η οικογένεια σου χάρτος της Ινδονησίας 15 με 35 δις ε, αμερικανικά δολάρια. Να, τι άλλο έχουμε. Να σου πω και κάποια άλλα παραδείγματα του τι γίνεται. Τα τροπικά δάση, Φιλιππίνες, ε, Μαλαισία, Ινδονησία δίνουν ευκαιρία στους ε, πολιτικούς να γίνουν πλουσιότεροι. Και αυτό έχει γίνει αντικείμενο και απεδείχθη ότι το εισόδημα από αυτά τα τροπικά δάση ε, ε τους, τους, τους, τους πλουτίζει και τους βοηθάει να καταστρέψουν τους κρατικούς θεσμούς. Και έτσι αυτές οι αντισώμενε χώρες που έχουν τόσο, τόσο κοιτάζοντα πετρελαίου γίνονται λιγότερο δημοκρατικές. Αν αυτό φαίνεται κακό υπάρχουν και χειρότερα διότι η φορολογική παράδειση, όχι μόνο δίνουν κάποιο κρυψώνα σε κάποιους να κρύψουν τα χρήματά τους αλλά αρνητικά επηρεάζουν τον τρόπο διακυβέρνησης των χωρών αυτών. Έχουμε 27 δε χώρες νοτίως της Σάχαρα στην Αφρική και την ώρα της μόνο 5 εξ αυτών είχαν προεδρία. Οι υπόλοιπε ήταν κοινοβουλευτικέ δημοκρατίες και τώρα που μιλάμε και 27 αυτές χώρες είχαν έχουν ε, γίνει προτρεβόμενες δημοκρατίες εκτός από τρεις. Τον Μαυρίκιο, την Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία και την Μποτσουάνα. Υπάρχει δε μακρύς κατάλογος ε, προέδρων οι οποίοι έχουν επεξαιρέσει το κοινωνικό χρήμα, το κοινωνικό πλούτο. Θα μπορούσα να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάλογο και να σας εξετάσω γιατί έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Όλοι αυτοί, Μουγκάμπε, αυτοί που σας είπα προηγουμένω. Αυτό είναι επομένω το φημισμένο παράδοξο των πλουσίων. right Αυτού του είδους η υπεξαίρεση που την, των, τον πόρων οδηγεί σε λιγότερη ανάπτυξη. Παρά το ότι αυτές οι χώρες έχουν, έχουν, έχουν ε, πρώτες ύλες, οδηγούνται όμως σε φτώχεια. Να το παράδοξο και γι' αυτό έχουμε αυτό το, αυτή τη φθήνουσα τάση. Όσο πιο πόρους έχεις τόσο λιγότερη ανάπτυξη έχεις. Όμως και η δική μου χώρα, και η δική μου χώρα η Νορβηγία τα πάει καλά. Άρα ποια είναι η διαφορά, γιατί αυτές οι χώρες είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές, ποια είναι η απάντηση. Ε, έχετε εδώ πέρα αυτές τις δύο φθήνουσες τάσεις και δείχνει ότι οι χώρες που έχουν σωστούς θεσμούς δεν επηρεάζονται από αυτό το παράδοξο του πλούτου. Δεν έχουν αυτή την ε, αρνητική σχέση μεταξύ ανάπτυξης και πόρων. Όμως αυτοί που κακεί την κυβέρνηση πάνε χειρότερα. Και είναι όλες οι κοινωνικές δημοκρατίες αυτές που τα πάνε καλά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν σωστοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και η φορολογική παράδοση που δίνουν τις ευκαιρίες στην άρχουσα τάξη τους δίνουν την ευκαιρία να μην εσωτερικεύσουν το κόστος των πράξεών τους. Διότι αν δεν είχαν αυτές τις κρυψώνες, τότε θα έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους στη χώρα τους και να έρθουν πρόσωπο πρόσωπο με τους συμπατριώτες τους. Η Δύση όμως υποστηρίζει τους πολιτικούς παραδείσους και θεωρεί ότι εντάξει αν δεν πληροφορίες αυτό θα λυθεί. Όμως φορολογικοί πάντα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τίποτα δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα. Άρα προτείνουμε το να γίνει μια διεθνή σύμβαση διαφάνειας και να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα επιλογή φαινόμενα σε εθνικό επίπεδο. Λέμε θέλουμε περισσότερα μέσα ούτως ώστε να μπορέσουμε να σταματήσει να σταματήσουν να πληρώνουν την ύφη για τις πολυεθνικές οι φτωχότεροι. Να υπάρξουν φορολογικά μέτρα και να υπάρχει ένα κέντρο για τα δημοσιονομικά διεθνές και για τη διεθνή φορολογία. Να ελέγχονται επίσης οι πολυεθνικές. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποια εταιρεία ανήκει σε ποια να μην πηγαίνουμε από θηγατρική σε θηγατρική, ούτως ώστε ο ισχυσμός του καθενός να είναι διάφανος. Αυτά όσον αφορά για τις πιο πλούσιες χώρες που τώρα λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουν τους φτωχότερους τώρα. Δεν θεωρούμε ότι είναι εδώ να έχουμε κάποιο άλμα. Το άλμα προόδου μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρξει βοήθεια προς τις ομένες χώρες να απαλλαγούν από τα παράσιτα που τις παραλύουν. Νομίζουμε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε κάτι για να άρουμε αυτό το τόσο βασικό φραγμό των φτωχότερων προς την πρόοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισηγήση σας, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο επόμενος ε, αγορητής θα είναι ο κύριος Μπέικερ της Global Financial Integrity. Σας ευχαριστώ. Ένας φιλόσοφος του Πανεπιστημίου Γιέλ Τόμας Πόγκη, και άλλος σημαντικός οικονομολόγος, το Βάνι Κόλλης και δύο Αμερικανοί, υπολογίζουν ότι περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι τον χρόνο πεθαίνουν από οικονομικές στερήσεις. Αν ο αριθμός αυτός είναι περίπου ακριβής ή περίπου τάξης μεγέθους, σημαίνει ότι σε αυτές τις τρεις ώρες ε, σήμερα το απόγευμα πρόκειται να πεθάνουν 6.000 άνθρωποι από στερήσεις ή από αιτίες οι οποίες προκύπτουν από τις στερήσεις αυτές. Η σκέψη αυτή μας αναγκάζει να θέσουμε ολόκληρη αυτή την εξίσωση της, ε, των οικονομικών παραγόντων επιτάπητος. Δεν έχουμε <clears throat> την πολυτέλεια να είμαστε επιλεκτικοί στα όσα θέλουμε να ε, εξετάσουμε ή όχι. Αυτή η ολόκληρη οικονομική εξίσωση για την ανάπτυξη, με όποιο τρόπο και να την εξετάσουμε, θα πρέπει να περιλαμβάνει το συνολικό κεφάλαιο των αναπτυσσόμενων χωρών, το κεφάλαιο που φεύγει από τις αναπτυσσόμενες χώρες και το τι μένει. Για να διατηρήσουμε αυτό το πιο ανοιχτό πνεύμα στην ανάλυση των θεμάτων αυτών, προσθέθηκε κάτι το νέο στην ατζέντα της παγκόσμιας οικονομικής ανάλυσης. Οι αρχικές ροές κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες θεωρούνται τώρα πια ε, σημαντικό μέρος της συνολικής οικονομικής εξίσωσης. Και η κίνηση αυτή έχει επιταχυνθεί τις ε, τελευταίες, ε, ε, τα τελευταία χρόνια. Το 2006 και το 2008 η Νορβηγία έκανε τρεις διασκέψεις κορυφής για να εξετάσει τα θέματα αυτά. Από τις διασκέψεις αυτές προέκυψε μια ομάδα ηθικών καθηκόντων για την οικονομική ακαιρεότητα με συμμετοχή 60 χωρών, μη κρατικών οργανώσεων και ιδρυμάτων που, αντιμετωπι... που εξετάζουν όλοι το σύνδεσμο μεταξύ των θεμάτων αυτών. Η Γερμανία έφτιαξε επίσης μια ε, ομάδα εργασίας. Η Ισπανία στέλνει στην ήρθε στην Προεδρία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα θέματα αυτά σε υψηλή προτεραιότητα. Και η Παγκόσμια Τράπεζα το Σεπτέμβριο διέθεσε δύο μέρες για να συζητήσει τα θέματα αυτά. Και μάλιστα και πριν από λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη έγινε πάλι η διάσκεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα θέματα αυτά είναι πλέον επιτάπητος είναι οι διατυπώσεις που κάναμε έχουν περιληφθεί στα ανακοινοθέντα των G8 και G20. Παρ' όλα αυτά, απογοητευτήκαμε από το ανακοινοθέν των Υπουργών Οικονομικών του G20 της προηγούμενης εβδομάδας που δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη υποσχέσεις που έχουν γίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εμείς στις δυτικές χώρες είμαστε υπεύθυνοι για την δημιουργία του συνολικού παγκόσμιου συστήματος που εξήγησε προηγουμένως ο καθηγητής Σέλντον που έχει μέσα και ε, φορολογικούς παραδείσους και κρυμμένες, εκατομμύρια κρυμμένες εταιρείες, ανώνυμες, ανώνυμους λογαριασμούς, ε, trust, ε, δραστηριότητες πλησίματος χρήματος, ψευδείς τιμές για το εμπόριο και τις διαμεθοριακές διακινήσεις, και αφήνει παράθυρα στους νόμους των δυτικών χωρών που διευκολύνουν τη διακίνηση των χρημάτων μέσα σε αυτό το σκιώδες οικονομικό σύστημα και εν τέλει καταλήγουν στις δικές μας οικονομίες. Η πληρέστερη ανάλυση αυτής της σκιώδους ε, παγκόσμιας οικονομίας είναι αυτή η εργασία που έχει γίνει από τον καθηγητή Σέλντον και τους συνεργάτες του. Εάν διαβάσετε την έκθεση του Tax Havens and Development, θα το βρείτε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα τους, θα καταλάβετε, θα καταλάβετε τι γίνεται στη διαδικασία αυτή. Πρόκειται για εξαιρετική εργασία. Στο πρόγραμμα μας για την ε, παγκόσμια οικονομική ακαιρεότητα αναγνωρίζουμε τη σημασία. Εγώ στο βιβλίο μου κάνω ένα υπολογισμό 500 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Το βιβλίο μου λέγεται «Η αχίλιος πτέρνα του καπιταλισμού». Πήραμε και έναν οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας με 30 ετή και πλέον πήρα, ο οποίος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει δύο, οικονομικές, δύο οικονομικούς τύπους, την ε, μέθοδο υπολείπων της Παγκόσμιας Τράπεζας και τις στατιστικές του IMF πράγματα που έχουν χρησιμοποιήσει οικονομολόγοι επί δεκαετίε. Εμεί χρησιμοποίησαμε τα μοντέλα αυτά πρώτοι για να βάλουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διαθεσή μα από ε, τις αναψώμενες χώρες, ισοζύγια πληρωμών κλπ. Η ανάλυση μα δείχνει περίπου 850 δισεκατομμύρια μέχρι ένα τρισεκατομμύριο τον χρόνο να εξαφανίζονται παρανόμω από τις ε, ε, αναπτυσσόμενε χώρε και όλα σχεδόν τα χρήματα αυτά καταλήγουν στι δικέ μα δυτικέ οικονομίε. Η Νορβηγία εξέτασε τις εκτιμήσεις αυτές που κάναμε πολύ προσεκτικά. Νομίζουμε ότι είναι και συντηρητικό ο υπολογισμό αυτό, διότι δεν περιλαμβάνει για παράδειγμα το λαθρεμπόριο, δεν ε, περιλαμβάνει τι ψευδεί αναγραφές τιμών για υπηρεσίε και τα άειλα αγαθά που είναι επίση ε, ένα τεράστιο μέρο τη εξίσωση, ούτε περιλαμβάνει και δεδομένα από ε, χώρες που εκπροσωπούν ωστόσο το 1 το τρίτο του ΑΕΠ της Αφρικής. Όπως λέει ο καθηγητής Σέλιον, αν εξετάσετε τα νούμερα αυτά, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια που φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και το συγκρίνεται με την ε, ενίσχυση που δίνονται για ένα εκατομμύριο που, θα δείτε ότι για κάθε ένα δολάριο που δίνουμε γενναιόδωρα βοήθεια στις αφρικανικές χώρες, λαμβάνουμε 10 δολάρια από αυτές. Στα 48 χρόνια μου εμπειρίας, 15 χρόνια παραμονή μου στην Αφρική, δεν είδα τίποτα άλλο να κάνει τέτοια ζημιά σε αναπτυσσόμενες χώρες όσο αυτή η μαζική έκροη παράνομων κεφαλαίων. Αδειάζει τους ε, φυσικούς και άλλους πόρους, ανοίγει τεράστια κενά ακυρώνει τις επενδύσεις, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και υπονομεύει το εμπόριο. Άλλο θέμα η οικονομία, άλλα τα εξωτερικά, άλλο το περιβάλλον. Μέσα στα οικονομικά λοιπόν τίποτε άλλο δεν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά σε αναπτυσσόμενες χώρες όσο αυτή η μαζική εκροή χρημάτων. Αυτό το παγκόσμιο σκιώδες οικονομικό σύστημα το οποίο διακινεί τα χρήματα αυτά είναι το πιο αποκρουστικό κεφάλαιο της παγκόσμιας οικονομίας από την ε, δουλεία και μετά. Κι όμως τα χρήματα αυτά είναι και η μεγαλύτερη πηγή ανάπτυξης για το μέλλον. Αν μπορέσουμε να περικόψουμε από τις ροές αυτές το 1 τέταρτο, το μισό ή το περισσότερο, θα πολλαπλασιάσουμε τα ωφέλη υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών για την μείωση της φτώχειας, για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς τα κόβεις τα ρεύματα αυτά ωστόσο. Μαθαίνω ότι η Επιτροπή σας πρόκειται να συμμετάσχει ε, μαζί με άλλες επιτροπές σε δύο συνεδριάσεις που θα τα συζητήσουν τα πράγματα αυτά. Τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να περικόψει κανείς τις ροές αυτές. Δεν θα πω σε αυτό όμως για την ώρα, αλλά θα σας ε, μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις. Ο στόχος είναι να περιοριστούν οι εκροές αυτές, όχι να ανακοπούν εντελώς. Γιατί για να ανακοπούν εντελώς χρειάζονται δρακόντια μέτρα. Περικοπή. Δεύτερο, αυτό μπορεί να γίνει με σχετικά μικρό αριθμό απλών μέτρων, εφόσον όμως αυτά ε, εφαρμοστούν με συνέπεια. Ο περιορισμός του φαινομένου δεν είναι και πυρηνική φυσική, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Βλέπω με ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με το θέμα αυτό με αυξανόμενο ενδιαφέρον και ρυθμό. Ηγετικό ρόλος για την προσπάθεια αυτή πρέπει να προέλθει από την Ευρώπη. Με την κυρία Ζολή, με την οποία έχω με μεγάλη χαρά συνεργαστεί στο παρελθόν, είναι εξαιρετική πρόεδρος για να σας ε, οδηγήσει στο μονοπάτι αυτό debo entender que el aplauso ha sido a ambos, al orador y a la presidenta. Eh, Α, φαντάζομαι και εκείνη χειροκροτήρα, όχι μόνο εσά. Πέτρο Δασκοντέλος είναι ο επόμενος ομιλητής. Έχετε 15 λεπτά. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε, είναι τιμή μου. Και όπως προείπα, τώρα Έχουμε την ε, ομάδα για τα εμβάσματα που συνδυάζει στη Ρώμη. Ε, συζητεί ακριβώς αυτό που συζητούμε και εμείς σήμερα. Το τι γίνεται με τις ροές των εμβασμάτων σε σχέση με την κρίση. Σε 15 μήνες θα προσπαθήσω να σας ε, δώσω μια γενική έποψη όσον αφορά αυτό το φαινόμενο, τα συμπεράσματα του τι γίνεται τώρα από πλευράς των αποτελεσμάτων της, του, του, του, του φαινομένου και επίσης πώς βλέπουμε τις εξελίξεις τα μέσα επόμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι το βλέπετε, αλλά αυτό που προβάλλεται στην διαφάνεια είναι ένας ορισμός. Ανεκαλύφθησαν ξανά τα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τελικά θα υπάρχει τόσο ενδιαφέρον. Είναι κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο το εμβάσμα. Όμω, εδώ εμπλέκονται και άλλα θέματα και άλλα συμφέροντα. Ε, δημόσιο τομέα, ο ιδιωτικό τομέα, η κοινότητα των πολιτών. Είναι ένα ανθρώπινο φαινόμενο, όμω τελικά πρόκειται περί χρημάτων και για να καταλάβουμε τι γίνεται σας δείχνω αυτό τον χάρτη. Πρόκειται για τις ροές των ε, εμβασμάτων προ τον αναπτυσσόμενο κόσμο μια εκτίμηση του 2006. Σήμερα είμαστε το 2009. Εκεί ε, έχουμε και 200 εκατομμύρια, τώρα μιλάμε για 218 δις. 200 τότε, 218 τώρα. And, uh, some, uh, some other studies, even though the correct... Και τα στοιχεία είναι από διάφορες πηγές και από δόσμια Τράπεζα, αλλά ε, αυτά είναι προσεγγιστικά γιατί πάρα πολλέ κεντρικέ τράπεζε δεν έχουν ιδέα ακριβώ περί του συνόλου τη της εικόνα. 300 δι λοιπόν έχουμε ε, παντού ε, λόγω τη κρίση. Σαν τζίρο βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, ιδίω στι αναπτυσσόμενε χώρε. Και για τι περισσότερε από αυτέ τι χώρε, τι αναπτυσσόμενε, βλέπετε ότι αυτή η ζωή του ξένου κεφαλαίου αντιπροσωπεύει περισσότερο από οτιδήποτε άλλη αρρωγή, ενίσχυση άμεση επένδυση, ιδίω τώρα σε, σε συγκυρία κρίση. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για την Αφρική. Όπου τα εμβάσματα, του στοχού προ του στοχότερου και γενιέ του είναι κάτι που υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη ροή. Δεν μπορούσατε να φανταστεί κανεί σε πολλέ φορέ δε. Έχουμε ε, Κάτι το οποίο ξεπερνάει τρεις φορές τις υπόλοιπε εισρωέ και εκροέ κεφαλαίων. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες ε, επίσης έχουμε τις, ε, τα την, την κορυφαία εισρωή. 60% πάνε σε, ε, στην Ήπεθρο, 25% του, ε, του, του ΑΕΠ είναι από τι εισρωέ, όπω η Σομαλία, το, το, το Πράσινο Ακροτήριο, Ερυθρία κλπ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, 200 δι και πρόκειται για ιδιωτικέ ροέ στην επόμενη πενταετία θα φτάσουμε τα 200 δις δολάρια τα οποία πρόκειται να εισρεύσουν στην Αφρική. Συζητούμε μόνο τώρα και προγραμματιζόμαστε για το ποιε είναι οι συνήθειε από, τις, ε, από τα εμβάσματα. Όταν λέμε να εννοούμε κόστο. Τα πάνε γιατί πριν από λίγα χρόνια θα έπρεπε ένα φτωχό μετανάστη να στείλει 200 δολάρια στην οικογένειά του και γι' αυτό θα έπρεπε να πληρώσει 20 με 25% προμήθεια. Και αυτό το κάνει κάθε μήνα. Δεν μπορεί να το κάνει όπω ε, εσεί και εμεί ε, όταν χρειάζεται να πάει να στείλει 1000 ευρώ. Δεν μπορούσε να το κάνει έτσι και θα μπορούσε να το κάνει ε, στο τέλος του μήνα αφού πληρωθεί και η προηγούμενη προμήθεια αυτά που σας είπα δεν υπήρχε άλλη λύση και και έχουμε διάφορες ε, εταιρείε που το κάνουν και καλά κάνουν δουλειά του όμως είχαν το μονοπόλιο, Ούτω ώστε να μπορούσαν να φτάσουν στι ε, υπηρεσίε τη υπαίθρου της μου της, της Κένιας και ε, χρέουν 25%. Τώρα μετά από 10 χρόνια το κόστος του εμβάσματο είναι κάτω από το 5%. Πάντα μιλάμε για την ύπεθρο τη Κένιας. Και ξέρετε πώς το κάνουν, όπως περισσότεροι από εμάς εδώ, με κομπιούτερ ή με κινητό. Έτσι για να καταλάβετε τη διαδρομή που κάναμε σε αυτή την δεκαετία. Και έτσι βρέθηκε αυτή η λύση για να στέλνουν τα βάζοντα στις οικογένειες. Τώρα, ο συμβή της κρίσης είναι το τι θα γίνει με αυτές τις ροές. Να σας, δείξω αυτόν τον χάρτη περισσότερα, αν σήμερα από ό,τι πρόπερση, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμα περισσότερα. Το είναι συνέπεια της μετανάστευσης. Συνέπεια της έλλειψης οικονομικών ευκαιριών. 200 εκατομμύρια και παραπάνω μεταναστεύουν τη σήμερα ημέρα, αφήνοντας την οικογένειά τους πίσω, πάνε και ζουν μια ζωή με γεμάτη θυσίες και δεν ξέρουν πότε θα ξαναγυρίσουν πίσω. Άρα στέλνουν συνεχώς στις οικογένειε τους. Στη ΣΥΠΑ ή στην Ευρώπη προσπαθούμε να εντάξουμε τους μετανάστες Ό,τι κάνουμε πάντως, αυτοί συνεχίζουν και στέλνουν τα λεφτά στις οικογένειές τους γιατί χρειάζεται να τα κάνουν. Πολλές από τις οικονομίες εκείνες, εάν κοβόντουσαν τα εμβάσματα, θα κατέρεαν. Και τώρα εδώ δεν μιλάμε για αναπτυξιακά ταμεία και δωρεές κυβερνητικές. Μιλάμε για κάτι που πηγαίνει από την τσέπη του μετανάστη στην άλλη τσέπη. Το 90% αυτών των χρημάτων πάνε στην κατανάλωση. Άρα βλέπετε πώς συνδέονται τα εμβάσματα με την παραγωγικότητα. Πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι ερωτήσει επομένως. βλέπετε ότι στην Αφρική έχουμε λόγω της κρίσης μείωση κατά 10%. Και το ίδιο για η Αμερική. Μεταξύ 6 και 10% είναι η συρρήκνωση αναχώρα κατά μέσο όρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών. Πάντως μιλούμε για πολλά χρήματα τα οποία χάθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Δεν τα παίρνουν πια οι οικογένειες. Και δεν μιλάμε για οικονομική κρίση, μιλάμε και για την τιμή των τροφίμων. Οπότε, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι κατά κάποιο τρόπο σε αναπτυσσόμενε χώρε. Στην συγγνώμη, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως λέγαμε τώρα συνδυάζει αυτή η ομάδα για τα εμβάσματα στη Ρώμη και φαντάζομαι περίπου τέτοια ώρα θα κλείνουν τη συνάντησή του ή και την, την, την εκδήλωση γενικότερα και το τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Μεγάλο ερωτηματικό πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση των ροών. Όλα θα εξαρτούν βέβαια και από τι ισοτιμίε, το συνάλλαγμα, το δολάριο. πάντω σε πολλέ περιπτώσει θεωρούμε ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση κατά το 6% και κατά το 2011 πάλι θα εξαρτηθεί από τις μεταναστευτικές ροές. Δεν νομίζουμε θα υπάρξει πτώση περαιτέρω. Όμως θα κάνει τη διαφορά το πώς θα εξελιχθούν οι ισοτιμίες. Οπότε τώρα η ουσιαστική προβληματική ακολουθεί. μια που το έμβασμα είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αφού μιλάμε για το κόστος της προμήθειας, θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος για το πώς τα εμβάσματα θα ωφελήσουν την ανάπτυξη. Άρα, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει κανείς είναι να δούμε το τι θα πρέπει να γίνει. δεν θα πρέπει φυσικά να υποκαταστήσουν τις αναπτυξιακέ προσπάθειες τις τέτοιες, τέτοιες Διότι λέμε 200 εκατομμύρια πάνε σε αυτούς γιατί δεν τους δώσουμε τότε αναψυχική βοήθεια. Όχι, είναι άλλη διάβλη είναι ιδιωτικέ ροέ. Δεν είναι η ίδια κατάληξη αυτών των χρημάτων. Αντιστοιχό μοντέλο για κάποια χώρα. Έχουμε θετικά και αρνητικά συμπεράσματα και συνέπειες από τα εμβάσματα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, εδώ έχετε μια μικρή εικόνα των όσων σας είπα. Είναι συνέπεια της μετανάστευσης είπαμε. Και βλέπετε ότι εάν δεν υπάρχει φαινόμενο μόχλευσης τότε έχουμε αποστέρεση του κόσμου στην Ήπεθρο από τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Φεύγουν και πάνε, ξέρω εγώ πάνε, ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, βέβαια το ελαττήριο και, το, η αιτία είναι ότι δεν υπάρχει τοπική οικονομική δραστηριότητα. Όμως μπορεί αυτός ο κύκλος να σπάσει με, με το, κάποιο φαινόμενο του μοχλού, Αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση έχουν περισσότερα εμβάσματα. Συρρήκνωση επίση της προμήθειας όπως προτείνει το G8. Οπότε θα έχουμε άλλα 200 δις τα οποία θα εκρέψουν προς εκείνες τις χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό που έγινε την τελευταία δεκαετία στη Λατινική Αμερική. Το πρόβλημα ήταν η παραπληροφόρηση. Δεν υπήρχε ούτε ανταγωνισμός. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πληροφορίε και δεν μιλάμε για 5 δις, αλλά για 16. 64 δις δολάρια που πήγανε στην Νότια Αμερική από τους μετανάστες του αγαπημένους τους. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού στην αγορά που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες και από τη μια άλλη πλευρά παρουσίασαν κάποιο πρόσωπο και έτσι μπόρεσαν να στείλουν περισσότερα χρήματα. Όμως, από και και σε αυτό το σημείο, θα πρέπει κανείς να δει το πώς θα έχει περισσότερες επιλογές ο μετανάστες. Όλοι είμαστε εδώ πέρα, έχουμε επιλογές διαφορετικές όσον αφορά το πορτοφόλι μας. Όμως, πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει. Όταν παίρνει το, ένταλ, το έμβασμα, ή τα βάζει στο στρώμα, τα κρύβει, ή πάει και τα ξοδεύει. Αυτό είναι που το κλειδί για το μέλλον. Πώς θα υπάρξουν ευκαιρίες. Είναι επίσης γνωστό ότι το ότι έχουμε τα μικροπιστωτικά ιδρύματα και άλλα φαινόμενα που σχετίζονται με το έμβασμα, αυτό είναι και θέμα του να μην κάνεις αναλφάβητος, το συμπίνει οικονομικά πραγματικά εκεί αν υπάρξει βελτίωση θα αλλάξει το πρόσωπο του κόσμου. Και έχουν αυτές τις προτάσεις του G8. Να, αυτές είναι οι προτάσεις. Οι συστάσεις που κατευθείαν ε, προέρχονται από την Τίνιδα που συνεδρίασε τελευταία φορά η ομάδα για τα εμβάσματα. Και ισχύουν βέβαια για όλο τον κόσμο, για τις εμψώμενες χώρες παντού. Η γνωστή ιστορία, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Κάτι το οποίο έχει εντυπωσιακή επίδραση στην ε, προμήθεια επί των ε, εμβασμάτων. Πώς να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλες οικονομικές υπηρεσίες οι εμπλεκόμενες στην αγορά. Μικροπιστωτικά ιδρύματα, τα διάφορα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να ληφθούν αυτά τα εμβάσματα και έτσι να υπάρξει περισσότερη δυνατότητα για τοπικές οικονομικές δραστηριότητες. Νέες τεχνολογίες που πραγματικά φέρνουν θαυματουργές αλλαγές και έτσι έφτασε στην τελευταία γωνιά της επέθρου το φαινόμενο και το τελευταίο είναι να υπάρχουν περισσότερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που να διατίθενται και στην Ήπεθρο. Να το φαινόμενο του υπομόχλειου. Γι' αυτό μιλάμε για 200 εκατομμύρια που έχουν τους αγαπημένους τους σε τέτοια μαξιμένα σημεία όπου εκεί υπάρχει ανάγκη για περισσότερο παραγωγικό τρόπο αξιοποίηση των εμβασμάτων. Υπάρχουν πάντοτε κάποια νομοθετικά πλαίσια και να, εδώ πέρα βλέπετε ε, τους ε, σύνδεσμους του, στο ίντερνετ. Αυτό είναι, αυτό αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες ε, ε, συγκεκριμένες συστάσεις. Ξέρω ότι ξεπέρασα το χρονικό όριο, συμπαθάτε με. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές, οι οποίοι τυχόν θέλουν να λάβουν το λόγο για να υποβάλουν ερώτημα για οποιαδήποτε από τι τρει εισηγήσει ακούσαμε. Ο κύριος Κάσμαρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσίαση αυτή για την λεύκανση των παρανομών προσόδων, τους φορολογικούς παραδείσους και απλώς θα συμφωνήσω κι εγώ ότι πρέπει να υπάρξει μια διεθνή σύμβαση για το θέμα αυτό. Είναι θέμα πλανητικό πλέον, όπω και οι κλιματικέ αλλαγέ. Δεν μπορούμε να το λύσουμε σε τοπικό επίπεδο. Η φορολογική παράδειση πρέπει να εξαλειφθούν ολοσχερός. Δεν μπορούμε να το λύσουμε σε μία χώρα μεμονωμένη. Το πρόβλημα όμως μιας διεθνούς σύμβασης θα ήταν ότι οι διαπραγματευτές θα δέχονταν πάρα πολλέ πιέσει και η ίδια η σύμβαση θα έπαιρνε πάρα πολύ καιρό μέχρι να κυρωθεί και να υλοποιηθεί. Έχουμε πολλέ συμβάσει. Αλλά ξέρετε πόσα χρόνια και δεκαετίε να περάσουν μέχρι τελικά να υλοποιηθούν οι συμβάσει αυτέ. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μια νομική βάση στο διεθνέ δίκαιο για να μπορέσουμε να το πετύχουμε, το στόχο αυτό τη σύμβαση. Αναφέρατε την έννοια τη ε, κατοικία, τη έντρας. Είναι κάτι που πολλέ ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν και κάποιε αφρικανικέ. Μπορεί κανεί να καταβάλει του φορού. μέσα σε 183 μέρες όταν είναι κάτοικος της χώρας. Οπότε αγοράζει το δικαίωμα να καταβάλει τους φόρους σε μια συγκεκριμένη χώρα εάν κατοικεί εκεί το μισό χρόνο ουσιαστικά. Εάν πρέπει κάποιος να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο για 183 μέρες, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί απλώς να είναι περαστικός, πρέπει να έχει μια επιχείρηση, να έχει κάποια φυσική παρουσία στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι μια ψεύτικη εταιρεία που απλώς να έχει την επιγραφή και το όνομα του φορολογουμένου. Θα έπρεπε λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή της έδρας και τη κατοικία και στους φορολογικούς παραδείσους για να τους εξαλείψουμε. Εάν οι εταιρείε έπρεπε να εδρεύουν σε μια συγκεκριμένη χώρα για μισή χρονιά τουλάχιστον, θα Βλέπαμε αν θα καταφεύγαν τόσο πολύ στους φορολογικούς παραδείσους στην Ιγυρία. Έχουμε 300 δις δολάρια από την πώληση φυσικού πετρελαίου. Αυτά τα κέρδη καθόλου δεν επενδύονται στην ίδια χώρα, στην ίδια τη χώρα, αλλά μεταφέρονται σε άλλες ε, σε άλλους προορισμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια λύση απλή, μια λύση που να δώσει αμέσως αποτελέσματα. Ευχαριστούμε η κυρία Ζολή. Νομίζω ότι σπανίως είχαμε τη δυνατότητα να δράσουμε τόσο αποτελεσματικώς για την ανάπτυξη παρεκτός από την περίπτωση αυτή ακριβώς των φορολογικών παραδείσων. Εδώ πραγματικά έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουμε την πραγματικότητα που μας περίγραψε η κυρία Τραωρέ και να τη συγκρίνουμε με την εκμετάλλευση των πρώτων υλών, την καταπολέμηση της αποξήλωσης, την ε, καταπολέμηση της, ε, των παράνομων χωματερών σε συνδυασμό με τους φορολογικούς παραδείσους. Ο καθένας εδώ θυμάστε τι έγινε στην ακτή του Ελεφαντοστού όπου απερίφθησαν τόσα τοξικά απόβλητα εξαιτίας της διαφθοράς του συστήματος της χώρας. Μιλάμε για μια εταιρεία που ήταν καταχωρημένη σε ευρωπαϊκή χώρα με φορολογικό καθεστώς που δεν απαιτούσε ε, ούτε να είναι εγγεγραμμένη σε μητρό, ούτε ελέγχους. Απαλλάχθηκε λοιπόν από τους ρυθμιστικούς ελέγχους. Μιλούσα για την τράφικ και την, ε, τις κατοχώρες εδώ σε αυτή την περίπτωση αλλά η φορολογική αυτή παράδειση υπάρχουν και η ύπαρξή τους είναι πραγματική, ε, πραγματικό αίτιο της υπεραλίευσης, της αποψήλωσης. Θα υπήρχαν πολύ λιγότερα τέτοια φαινόμενα, αν δεν μπορούσε κανείς να ξεπλύνει το βρώμικο αυτό χρήμα στους φορολογικούς παραδείσους. Έχω λοιπόν ένα ερώτημα να θέσω στον καθηγητή Σέρντρουπ θεωρείτε ότι τα μέτρα που ο ΣΑ προτείνει μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των φορολικών παραδείσων και το πρόβλημα που αυτοί οι παράδεισοι εκπροσωπούν για τις ερωτησόμενες χώρες. Ευχαριστούμε, κυρία Ζολή. Η κυρία Εολίνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλες και όλους τους παρεμβάντες. Εξαιρετικά ενδιαφέρον απόγευμα και μακάρι να ήταν εδώ και περισσότεροι ευρωβουλευτές. Ελπίζω η έκθεση του κυρίου Σέρντερουπ, του καθηγητού Σέρντερουπ, να διανεμηθεί σε όλους τους βουλευτές, γιατί θα είναι μεγάλη ωφέλεια από την αναγνωσή της. Με τρόπο διαυγή φάνηκε καθαρά, μας δείξατε καθαρά, ότι η ίδια ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων οδηγεί στην αποδυνάμωση των θεσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες. δίνουν όθηση σε δυνάμεις που υπονομεύουν τους θεσμούς. Όπως είπε η ίδια η κυρία Τραωρέ, η ρίζα του κακού, του κακού στην Αφρική σήμερα είναι ιδίω η διαφθορά. Πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους. Και με τον τρόπο αυτό ληστεύουν τους λαούς. Τους στερούν τα πλούτη, τα οποία δικαιωματικά τους ανήκουν. Ακούστηκαν ποσά πραγματικά ηλικιώδη. Ακούστηκε επίσης ότι τα κονδύλια ρέουν, εκραίουν, φεύγουν από τις αναψώμενες χώρες. Τα λέει αυτά η έκθεση. τα μισά από τα κονδύλια αυτά είναι, ε, ε, μάλλον θα ήθελα να, το πω διαφορετικά. Θα ήθελα να γνωρίσω ποια είναι τα ποσοστά, πώς χωρίζονται δηλαδή τα κονδύλια αυτά ανά ε, περιοχή του κόσμου, από την Ασία, την Αφρική κτλ. Η Φραντσέσκα Κέλλερ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες και όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Ερώτηση προς τον καθηγητή Σιέρντερουπ. Είπατε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα πράξεις φορολογικών εσόδων. Ωστόσο, πώ θα γίνει αυτό στην πράξη. Γιατί είπατε ταυτόχρονα ότι οι ηγεσίε του χρησιμοποιούν φορολογικού φορολογικούς παραδείσους. Ε, πώς, εν πάση περιπτώσει, να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει από ευρωβουλευτέ, θα δώσω το λόγο στου εισηγητέ και εάν επιθυμούν να σχολιάσουν και κάτι άλλο από αυτά που άκουσαν. Πολύ ευχαριστώ. Εσείς κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα, τις, θα σας απαντήσω ως εξής. Στην Δύση μαθαίνουμε στα παιδιά μας, τουλάχιστον στη Δύση, μαθαίνουμε τα παιδιά μας ότι αν δουλεύσουν σκληρά θα τα καταφέρουν και καλά. Διατηρώντας, διατηρώντας ωστόσο τους φορολογικούς παραδείσους, αυτό που διδάσκουμε στις ηγετικές ε, τάξεις ορισμένων χωρών είναι ότι εάν κλέψουν θα περάσουν καλά. Η ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων είναι ντροπή για όλους μας. Η φορολογική παράδοση, η παράδειση συγγνώμη, σκοτώνουν κόσμο στι αναπτυσσόμενες χώρες. και ε, πραγματικά δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα ευφυής για να βρει μέτρα για να ε, καταργήσει τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά πώς αντιμετωπίζεις αυτούς οι οποίοι έχουν τα συμφέροντα στους φορολογικούς παραδείσους. Έρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Ζολή. Εάν τα μέτρα που προτείνει ο ΩΣΑ ο, θα λύσουν τα προβλήματα των φορολογικών παραδείσων. Και η απάντησή μου είναι ένα μεγάλο όχι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν στον πυρήνα του προβλήματος. Η φορολογική παράδοση εν συνειδήσει πάνε να πλήξουν τις φορολογικές βάσεις των άλλων χωρών. Προσφέροντας και το απόρριτο των λογαριασμών, ώστε οποιοδήποτε κλέψει να πάει να τα βάλει εκεί, σε αυτούς. Και έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση. Προτείναμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια των χωρών και με φορολογικά έσοδα. Αλλά αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία γιατί το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν οι ακροές. Η πρώτη προτεραιότητα είπε και η Νορβηγική Επιτροπή θα είναι να μην επιτρέπονται οι παράνομε δραστηριότητε των φορολογικών παραδείσεων. Αν επιτύχουμε σε αυτό τότε θα έχουμε και πρόοδο και στα άλλα ε, τμήματα. Τέλο, ε, χαμηλά ποσοστά είπατε για την Αφρική. Μα η Αφρική είναι φτωχότερη από την Ασία. Γι' αυτό και τα ποσοστά για την Ασία των νεκρών κεφαλαίων είναι υψηλότερα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο μεγάλο και ίσω και μεγαλύτερο στην Αφρική από ό,τι στι άλλε χώρε. Αυτό που τονίζω είναι η αρχή την οποία όλοι αντιμετωπίζουμε, ότι εάν κάνεις κάτι το οποίο βλάπτει άλλους, θα πρέπει ίσως ο να υποστείς τις ευθύνες. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που λέμε επιτρέποντας να συνεχίζουν να, υπάρχονται, να υπάρχουν οι φορολογικοί παράδεισοι είναι ότι τους προσφέρουμε ατιμορρησία σε αυτούς τους διεφθαρμένους ηγέτες. Παράνομε ροές κεφαλαίων μέσω φορολογικών παραδείσων. Αν δεν τα ανακόψουμε αυτά, δεν πρόκειται να επιτελεστεί πρόοδος. Είπατε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, κύριε Κάσμαρεκ, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μακροχρόνιε διαπραγματεύσει. Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι οι χώρες, οι χώρες αυτές πάνω δεν πρέπει να ε, προχωρήσουν σε δράσεις. Ήδη ο ε, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει εκδώσει σχετικά ε, ψηφίσματα από το 1977 και χρειάστηκαν άλλα 20 χρόνια για να περάσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλοί στην Αμερική είχαν ανησυχήσει ότι θα χάσουν ανταγωνιστικότητα. Δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δυνατότητα οι ίδιε οι χώρε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Η Νορβηγία εξετάζει όχι μόνο ε, το ενδεχόμενο να υπογραφεί μια συνθήκη για την διαφάνεια, αλλά και τι μπορεί να κάνει και η ίδια. Τη κυρία Ζολή η ερώτηση για τον ΟΣΑ, τη διαδικασία του ΟΣΑ. Όπω γνωρίζετε, ο ΟΣΑ τονίζει, η ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή δημοσιονομικών φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των χωρών. Και ε, έχουμε φτάσει περίπου στις 120-130 ε, συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Εάν πάρετε 200 ε, φορολογικές δικαιοδοσίες που πρέπει να προβούν σε ανταλλαγή με άλλες 200, φτάνετε σε 4.000 συμφωνίες. Ε, αυτό που εννοώ είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά. Το συζητήσαμε και με τους αξιωματούχους του ΟΣΑ και νομίζω ότι ανεγνώρισαν την αλήθεια αυτά, ότι, αυτή. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσει κανείς πια και την και ε, την, ε, τις απλές διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Λόβενς. Για τη ρίζα του κακού δεν συμφωνώ που είναι η διαφθορά για τις διαμεθοριακές, διαμεθοριακές ροές ε, παράνομων κεφαλαίων. Όχι αυτά που μένουν μέσα στην ίδια τη χώρα. Συνολικά, παγκόσμια δηλαδή, ε, τα έσοδα από, ε, από λαδώματα όπως λέμε, είναι περίπου 3% ναι. και τα ε, έσοδα από ε, φορολογικούς παραδείσους είναι 66% περίπου των όλων κεφαλαίων που διακινούνται ε, παράνομα. Τώρα, ότι οι ηγετικές ελίτ εποφελούνται από τους φορολογικούς παραδείσους, ναι, αλλά μην ξεχνούμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τους φορολογικούς παραδείσους με αναγραφή ψευδών τιμών ε, στο εμπόριο με ε, άλλα ποικίλα τεχνάσματα τα οποία είναι συνήθις πρακτική των ε, μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων με στόχο να αποφυγούν την πληρωμή σε άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να φορτώσουμε μοναχά στι αναπτυσσόμενες χώρες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να είναι μια διμερής προσπάθεια. Για το ίδιο θέμα, να έρθω για να σας πω δύο θετικά πράγματα για τους Αφρικανούς μετανάστες. Διότι, παρά τόσα λέμε για αυτέ τις ροέ κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάνουν ό,τι μπορούν τόσο στη δική τους να πάρουν τα χρήματα που πρέπει. Και θρησκευτικά τα λατήρια πολλές φορές. Υπάρχει και αυτή η πτυχή. Πολύ σημαντική πτυχή αυτή. Το τι προσπάθειες κατάβαλαν τώρα κάτι άλλο για τα εμβάσματα. Κάτι το οποίο πολλές φορές αμφισβητείται. Το θέμα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ίσως ε, δεν είναι σαφές αυτό το οποίο είπαμε. Είπαμε ότι πολλές φορές υπάρχει συνδυασμός εμβάσματος με ξέπλυμα. Όμως για αυτούς που το κάνουν είναι η χειρότερη μέθοδος. Γιατί θα πρέπει χιλιάδες άτομα να εμπλακούν και από τις δύο πλευρές για να το κάνουν τη δουλειά. Διότι πάντοτε τα ποσά είναι μικρά. Και όσο προχωρεί η τεχνολογία αυτό γίνεται δυσχερέστερο. Άρα, από αυτή τη πλευρά δεν επηρεάζουν και πολύ τα πράγματα, τα εμβάσματα. May I a point, um, uh, Και εγώ θα έρθω να συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί όσον αφορά αυτές τις, ε, αυτή τη φυγή, διαρροή κεφαλαίων, δεν, δεν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τα εμβάσματα. Είναι άλλο. Η, η, κροή, η, η κεφαλαιων κεφαλαίων είναι 80-90% που ε, βγαίνουν και ξαναμπαίνουν τελικά διάφορους τρόπους στην χώρα προέλευσης. Απλώς να προσθέσω, λέει κυρία Τραωρέ, ότι από δικής μου πλευράς από τις δικές μας χώρες μπορούμε να αποθαρρύνουμε τους ε, απαταιώνες, τους κλέφτες εάν τα θύματα ανακτήσουν, απο, αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι τελικά όλες αυτές οι πληροφορίες κυκλοφορούν μεταξύ των μοιημένων. Οι Αφρικανοί που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, εάν ήξερε το τι γίνεται θα, θα ήταν μια, μια ψηφοφόρος που δεν είναι τώρα. Τώρα είναι ε, μέλος της Αγέλης. Μόνη της κάνει το τόντο και Και θα καταλήξει να πάει να ψηφίσει τον ίδιο. Τον ίδιο υποψήφιο ο οποίος θα γίνει ακόμα πλουσιότερος. Ο οποίος μετά θα, θα, θα ρίξει περισσότερο χρήμα, ώστε να ξαναεκλεγεί. Αυτό που σας για τη δημοκρατία στην Αφρική. Όμως αυτό που με ενοχλεί είναι ότι η Ευρώπη προσέχει περισσότερο τα τεχνικά, τις τεχνικές πλευρές, αν υπάρχει διαφάνεια κλπ. Όμως, όσον αφορά τις γυναίκες, όσον αφορά τους μετανάστες, σας διαβεβαιώ ότι μέσα σε πέντε χρόνια θα δείτε μια ριζική αλλαγή. Ε, muchas gracias. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ με γνώση, με σοφία ε, συμμετέσχουν ε, όλοι όσους καλέσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όσον αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης επί των απτυσσομένων χωρών. Οπότε και θα πρέπει επομένως και πάλι πάρα πολύ θερμά να τους ευχαριστήσουμε και όταν έρθει η ώρα να κάνουμε το σχέδιο κειμένου μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο ακούσαμε. Και τώρα κύριε Ζωλή, επίσης, ε, για άλλη μια φορά θα συνεχίσει την ε, άσκηση της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωλή. και τώρα θα, για να δούμε τι άλλα θέματα έχουμε όσον αφορά τις, τα αποτελέσματα της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης επί των αναπτυσσομένων χωρών. Και κάτσουμε να δούμε τι έγινε με την έκθεση την οποία ε, ετοίμασε ο κύριος Γκερένα. Έχετε το ρόλο κύριε Γκερένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια πρώτη προσέγγιση ε, όσον αφορά την έκθεσή μου. Όπως είπαμε πρόκειται για ένα σχέδιο κειμένου το οποίο θα το ξαναδούμε στην επόμενη συνεδρία του 2007 ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση τα αποτελέσματα ξεκινήσαν το 2008, αλλά έγιναν ακόμα πιο σοβαρά μετά από την κρίση της εταιρεία Lehman Brothers που βγήκε μετά από ένα χρόνο. Οπότε με το που βγήκαν από την οικονομική κρίση κάποιες χώρες αμέσως διαπιστώθηκαν ε, κάποια φαινόμενα. Πρώτα πρώτα ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν αποτελούν την αιτία της κρίσης. Δεν ξεκίνησε από εκεί η κρίση. Οι χώρες αυτές όμως υφίστανται τις πιο καταστροφικές συνέπειες του φαινομένου. Δεύτερο πράγμα το οποίο ανεφάνει είναι ότι είναι χρηματοπιστωτική αυτή η κρίση που στην αρχή λέγεται ότι δεν θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες μια που δεν είναι ενταγμένες πραγματικά ε, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όμως Φέτος η κρίση αυτή χτύπησε με καταστροφικό τρόπο. Οικονομικά, κοινωνικά, ε, νηπτυσιακά και ανθρωπιστικά τις χώρες εκείνες. Τρίτο πράγμα το οποίο προέκυψε είναι ότι οι αντισόμενες χώρες υποφέρουν από αυτή την κρίση σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητα. Υπάρχει λιγότερη οικονομική ανάπτυξη. Έχουν χειρότερο αριθμό απασχόλησης. Έχουν πέσει οι τιμές των πρώτων τους υλών συρρυκνώθηκε η παραγωγική δραστηριότητα, έχουν λιγότερη πρόσβαση σε ε, δανεισμό, ε, με προσφυγή στις διεθνείς τράπεζες, έχουν τώρα ε, έχουν λιγότερες επενδύσεις από το εξωτερικό και είναι λιγότερο, όπως ακούσαμε, τα εμβάσματα από τους μετανάστες. Μια που οι δωρητές επίσης προσπαθούν να ρίξουν τα χρήματά στην ανάπτυξη και σταμάτησαν να τους δίνουν χρήματα. Επίσης, από πλευράς ε, δημόσιου τομέα ε, έχουμε κάποια σχέδια ε, ανασυγκρότησης, συστήματα, συστήματα για την ρευστότητα και 25 προς 1 είναι ο λόγος του πόσο ρίχνονται κεφάλαια στις αναπτυχημένες χώρε σε σχέση με τι αναπτυσσόμενε. Οπότε, βγαίνουν σιγά σιγά από την κρίση οι αναπτυχμένες χώρες, αλλά οι αναπτυσσόμενε ακόμα ε, υφίστανται τις επώδυνες συνέπειε της κρίσης. Για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, η κρίση αυτή θα αποτελεί μία μικρή διακοπή σε μία διαρκή πορεία ευημερία. Ενώ στι αναπτυσσόμενε χώρε θα πρόκειται για έναν γκρεμό ε, έναν γκρεμό στον οποίο θα, θα κινδυνεύουν να γκρεμιστούν οι όποιε πρόοδοι σημειώθηκαν στην πορεία του κατά τη δυστυχία και κατά τη φτώχεια. Αυτό που θέλω να κάνουμε ε, στην έκθεση δεν είναι το να κάτσουμε να κάνουμε μια απλή καταγραφή. Δεν θέλουμε απλώ να κάτσουμε να καταγράψουμε ποιε είναι οι συνέπειε τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αντιθέτω, αυτό το οποίο θέλω να κάνω με την έκθεση είναι να απευθύνω έκκληση στην ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν δράση όσον αφορά αυτή την πραγματικότητα. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου που να μπορέσει να ε, καταστήσει πραγματικότητα μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Άρα τώρα χρειάζονται απαντήσεις ε, τώρα ε, του χρόνου, το 2010. Το 2009 και το 2010. Η διαπάντηση δεν είναι δυνατόν να αποτελείται από κάποια εμβαλωματικά, απομονωμένα, μεμονωμένα μέτρα όσο και αν αυτά μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει μια δέσμη αποφάσεων που θα δώσουν μια όθηση να προέρχεται από τα θεσμικά όργανα, από τα κράτη-μέλη ε, και θα πρέπει να καλύπτονται τα εξή. Πρώτον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις όσον αφορά την η βοήθεια. 56. Ε, το είναι πολύ λιγότερο το με αυτά το οποίο δεν σχέση με το ΕΕ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος το να, το να η βοήθεια ε, προς τις αντισόμενες χώρες. Άλλη, άλλη, άλλη, άλλο πράγμα πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει οι χώρες αυτές να βοηθούν από νέους πόρους, νέες, νέες πηγές. Ε, χρημάτων. Ας πούμε λέγαμε για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Άρα θα πρέπει με αυτά τα φορολογικά μέτρα να πάρουμε κάποια χρήματα με τα οποία, τα οποία να τα ρίξουμε σε αυτό το διεθνές σύστημα. Να γίνει αναψιακή βοήθεια, να υπάρξει επομένως να υπάρξουν νέοι πόροι. Γιατί κάποιες χώρες, η Γαλλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Σενεγάλη, Αυστρία, Χιλή, Νορβηγία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Νομένο Βασίλειο και Ισπανία συνεκρότησαν μια task force ούτως ώστε να δουν κατά πόσον αυτός ο φόρος επί των ε, συναλλαγών μπορεί να είναι κάτι το βιώσιμο ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα φορολογικά μέτρα, τα σχετικά επίσημα με το δεξιό του άνθρακο, τα σχετικά τα φορολογικά μέτρα για τι μεταφορέ, ούτω ώστε να μπορέσουμε έτσι να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματο σύμφωνα με την αρχή ότι ο Ριπένο πληρώνει. Αποφάσισαν οι Γερμανοί ο φόρο του διοξιδίου να πάει σε ψυχικά προγράμματα. Δηλαδή η Ισπανία θέλει έτσι να κάνει κάποιο είδου ε, εθελουσία φορολογία επί των αεροπορικών εισιτηρίων. Είδαμε τι σημασία έχουν τα εμβάσματα σε σχέση με το έπτον χρόνο εκείνο, άρα θα πρέπει να μην υπάρχει ούτε στη μία ούτε στην άλλη χώρα ε, επιβάρυνση αυτών των εμβασμάτων. Και να υπάρξει μείωση, μείωση κατά το ίμιση των, των προμηθειών των εμβασμάτων. Τα δε προγράμματα τα αναπτυξιακά θα πρέπει να είναι τέτοια που τις αποφάσεις σας λαμβάνει από τις όμορες χώρες. Aid for Trade. Και να υπάρξουν προγράμματα που να δημιουργήσουν υποδομές. Να βοηθηθούν οι μεταφορές που είναι ε, στοιχείο που προσδίδει δυναμισμό ή στην τοπική οικονομία. Όπως είδαμε και σήμερα, πάμε προς αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού. Έτσι, θα έχουμε πρόοδο όσον αφορά τις οικονομικές εταιρικές σχέσει, ιδίω για τι χώρε ΑΚΕ. Πέμπτον, να καταπολεμηθούν η φορολογική παράδειση. Κάτι το οποίο το οποίο το ακούσαμε. Ακούσαμε και για την Νορβηγία. Νορβηγία, Χιλία, Γερμανία και Ισπανία επίση τώρα συνεκρότησαν μια task force για να καταπολύσουν του παραδείσου. Επίση, κατά έκτον θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόριο όσον αφορά τη, τα, τα πολυμερή θεσμικά όργανα. Γιατί πολλοί από του σήμερα ομιλήσαντες είπαν ότι για να υπάρξει καλή, σωστή διαχείριση θα έχουμε ε, λιγότερη φτώχεια, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερο άμεσο σχετισμό μεταξύ τη προσπάθεια τη αναπτυξιακή και τη ύπαρξη, τη ωφέλειά αυτή τη προσπάθεια από τον πολίτη. Τέτοιου είδους ε, διαχείριση, διακυβέρνηση θα πρέπει να αφορά τι χώρε, αλλά θα πρέπει να αφορά και του πολυμερεί οργανισμού, του διεθνεί πολυμερείς οργανισμού και θα πρέπει οι χώρες αυτές να εμπλακούν με αυτά τα πολυμερή όργανα τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Φερρυπίν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να καταφέρουμε του χρόνου να γίνει αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας και επίσης του χρόνου να κάνουμε κάτι όσον αφορά τη δόνωση της στόχης. Το G20 ξεκάθαρα να τοποθετηθεί και να εφαρμόσει άμεσα ό,τι αποφασίσει ούτως ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους της χιλιετίας. Εν κατακλείδη θα πρέπει η Ντόχα να αποτελέσει μια ευκαιρία ούτως ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορέσουν να πετύχουν αυτά τα οποία μας είπε η καθηγήτρια Τραωρέ. Επανειλημμένα ότι δηλαδή δεν πρόκειται για λύση που προκύπτει από τη, τη λύπηση προς, τον, ε, προς τις χώρες που υποφέρουν από την φτώχεια και από όλα αυτά θα πρέπει κανείς να τις στηρίξει, να τους δώσει ευκαιρίες στο εμπόριο, στην οικονομική ανάπτυξη, ε, επί τη βάση των δικών τους προσπαθειών και των δικών τους δυνατοτήτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο για την πολύ εύστοχη αποτίμηση της κατάστασης ως ηγητής. Νομίζω είναι σημαντικό όταν κοιτάζουμε τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις αναπτυσσόμενες χώρες μαζί με την αναπτυξιακή βοήθεια. Να διαρωτώμεθα τι θα κάνουμε εμείς ως κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Ζητάμε πολλέ φορέ από άλλου να αναλάβουν δράση, αλλά σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δούμε εμεί τη δράση που μπορούμε να αναλάβουμε. σω επαναλάβω κάτι που έχει ξαναεποθεί εδώ, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη κάποιε βασικέ αρχέ. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει στο ΑΕΠ τους να, το, να παραμείνουν στη δέσμευση του 7% του ΑΕΠ τους και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας για τους στόχους της χιλιετίας και να τους επιδιώξουμε σαν να είναι στόχοι εφικτοί. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως ανεξάρτητα κράτη. Τα, το κόστος των ε, εμβασμάτων Είναι σαφές ότι μας απασχολεί, γιατί το κέρδος, τα κέρδη που προέρχονται από την αποστολή των εμβασμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι παράλογα. Η... Το πλαίσιο του ΟΗΕ και η δέσμευση κονδυλίων από τα κάτι μέλη για τους σκοπούς του ΟΗΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για όλους αποτελούν όλα αυτά ένα μέρος, ένα μικρό ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι μια μικρή συμβολή και θα πρέπει τα οικονομικά, οι υπεύθυνοι των οικονομικών των κατώμελών να το έχουν αυτό υπόψη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τους φόρους για τις οικονομικές συναλλαγές. Κάποιες χώρες αυτή την προσέγγιση είναι πιο προεδευτικές όπως η δική μου και η Ισπανία αλλά παρά την απογευματινή μας συζήτηση μην ξεχνάμε τα όσα υπόθηκαν τη μεταρρύθμιση των ε, καταστατικών για τους φορολογικούς παραδείσους τα ποσά που αυτή τη στιγμή διαφεύγουν σε αυτούς τους παραδείσους δεν θα πρέπει να μένουν εκεί. Θα πρέπει να τα πάρουμε από αυτούς τους παραδείσους, να τα φέρουμε πίσω. Είπατε για απληστία. Ναι, θα πρέπει καμία χώρα και να μην βρίσκεται σε δυσμενείς όρους σε σχέση με τις, σχέσεις, με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Και για τον εκπρόσωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου να πω ότι σαφώ πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χθε το συζητήσαμε μόλι. Ναι, επενδυτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Συμφωνούμε λοιπόν ότι και η Παγκόσμια Τράπεζα και το IMF πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Και πρόεδρε, χωρί καμία ειρωνία, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εξωτερικέ μα δράσει και οι πολιτικέ εξωτερικέ στηρίζουν του αναπτυξιακού μα στόχου και όχι αντίστροφα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουν το λόγο. No. Okay. Then we... Ωραία. Ίσως τότε να είχαμε κάποια καταληκτικά σχόλια από τον κύριο Γκερέρο. Δύο παρατηρήσεις θέλω να πω για να κατελήσω κάπου. Πρώτα πρώτα όσον αφορά την Κομισιόν και κάτι σε σχέση με όσο είπε ο κύριος Κάσμαν. Ελπίζω ότι όταν η έκθεση την να ολοκληρωθεί, να είναι πιο θετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όπως είπατε θέλουμε το Κοινοβούλιο να εξωθήσει την Επιτροπή να θεσπίσει κάποια μέτρα τα οποία να είναι χρήσιμα, ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε τις συνέπειες της ε, κρίσης για τις αντισωμένες χώρες. Δεν μπορούμε εμείς να θεσπίσουμε κάποια μέτρα ούτως ώστε οι χώρες αυτές κάτι να κάνουν. Στην επόμενη συνάντησή μας ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πιο θετική όσον αφορά τις προτάσεις μας. Για αυτό τώρα που είπε ο συνάδελφος Κάσμαν θέλω να σας ε, επισημάνω ότι σήμερα μπροστά μας ξανοίγονται κάποιες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να λάβουμε κάποιες ε, αποφάσεις που εάν δεν τις λάβουμε πρόκειται τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα. Τώρα έχουμε κάποια ευαισθησία, έχουμε κάποια ανησυχία, έχουμε κάποια δυνατότητα αντίδρασης. Όμως, σε λίγους μήνες, σε ένα-δύο χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν Ε, δεν θα υπάρχει το πρόβλημα για τις αντισόμενες ώρες. Και, όπως είπαμε, ε, σε σχέση με όσο είπε ο κύριος Κάσον, τις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε μάρτυρες ανησυχητικών εκδηλώσεων σε σχέση με αυτά που τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Έχουμε τη συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ, τον κύριο Μπράουν, για αυτό το, τον φόρο των συναλλαγών που θεωρήθηκε ως μορφή ενισχύσεως. Όχι σαν πηγή εισόδων για να υποστηρίξουμε τις χώρες εκείνες. Κάτι άλλο επίσης σαν σύγκομνη σχετικό είναι ότι καθώς πλησιάζει η Κοπενχάγη απομακρύνεται η λύση της Κοπενχάγης. Δηλαδή οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, αυτές που θα πρέπει να δεσμευτούν στην Κοπενχάγη και άλλες χώρες που αναδύονται τώρα, κάποιες χώρες που έχουν σημαντικές εκπομπές θερμοκηπίου αρχίζουν να είναι πιο διδακτικές σε σχέση με οτιδήποτε μέτρο και κίνηση που θα σήμαινε δαπάνες και κόστος οικονομικό. Εμείς από αυτή τη θέση έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει οι αναπτυγμένες χώρες να βοηθήσουν τις σε σχέση με τις δεμενείς συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Για προσαρμογή και για μετρίαση των συνεπειών αυτών. Πρόκειται επομένως για μια συγκυρία όπου έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Και θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα από κοινού τώρα να προσπαθήσουμε μαζί, γιατί τώρα ανοίγεται αυτό το παράθυρο στην ελπίδα. Και τώρα να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις της ε, συνεδρίασης των συντονιστών σήμερα το πρωί. Σε ό,τι αφορά τον διορισμό εισηγητών και εισηγητριών για γνωμοδότηση, αποφασίσαμε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, έκθεση πρωτοβουλίας, για την εντολή μετά μάλιστα τη χθεσινή συζήτηση με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Φίλιπ Μεστάτ, ε, θα ετοιμάσουμε μια έκθεση πρωτοβουλία για τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον τομέα τη συνεργασία για την ανάπτυξη και εν ώψη τη ενδιάμεση αναθεώρηση τη εντολή τη τράπεζα αυτή. Σε ό,τι αφορά τι γνωμοδοτήσει, η γνωμοδότηση για την ε, απαλλαγή του 2008 θα συνταχθεί από το ΕΛΚ Επίση, θα συνταχθεί γνωμοδότηση για λογαριασμό τη Ευρω... ΑΦΕΤ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική για μια συνεργασία μεταξύ διεθνών φορέων και θέλουμε να συνεργαστεί στη διαδικασία αυτή και η αρμόδια επιτροπή. Για τι κοινοβουλευτικέ ερωτήσει, ο Επίτροπο που θα αναλάβει την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξική βοήθεια εδώ το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται για την ακρόαση των ε, διορισμένων υποτρόπων και εφόσον οργανωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται για το τέλο αυτή τη εβδομάδα. Σημειώνουμε ότι μέχρι το τέλο του μήνα πολλά είναι τα μέλη μα που θα συμμετάσχουν στην ισότιμη, στη μεκτή κοινοβουλευτική επιτροπή τη στην Αγγόλα και η ακρόαση για τον μελλοντικό επίτροπο ορίστηκε τις 25 Νοεμβρίου μεταξύ 8 και 8.30 το βράδυ. Ένα ερωτηματολόγιο γραπτό θα ετοιμαστεί, όπως αποφασίσε η διάσκεψη των Προέδρων, για να κάνουμε με όλους τους επιτρόπους, και θα δοθεί έμφαση σε πέντε θέματα προτεραιότητας, για τα οποία οι Επίτροποι θα κληθούν να αναφέρουν τις νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που σκοπεύουν να, να προβλέψουν για την υλοποίηση των καθηκόντων του. Οι συντονιστέ συμφώνησαν για τι πέντε ακόλουθε προτεραιότητε. Θα τι διαβάσω στα αγγλικά, διότι δεν είχαμε το χρόνο να τι μεταφράσουμε. Επιδίωξη των στόχων τη χιλιετία ω το 2015 και υλοποίηση τη δήλωση τη χιλιετία και ιδιαίτερω τη διατάξει και δεσμεύσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καλή διακυβέρνηση και το κράτο δικαίου. Καθώ και διασφάλιση το ε, υπάρχοντο ρυθμό για την αναπτυξιακή βοήθεια μετά το 2015 βάση της αποτίμησης των επιτευγμάτων και των έλλειμμάτων από την ε, ως τώρα αναπτυξιακή συνεργασία. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της ένδυας, την επισητιστική ασφάλεια, την περιβαλλοντική ανάπτυξη και την ε, ενίσχυση του κοινωνικού ιστοτών αναπτυσσόμενων χωρών συμπεριλαμβανομένων τη διεθνού διακυβέρνηση που θα πρέπει να λάβει υπόψη τη θέση των αναπτυσσόμενων χωρών και να μην γίνει εργαλείο για άλλε εξωτερικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των αξιών ε, της ιδιοκτησίας, της αξιοπρέπειας, της εταιρικής σχέσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ευθυγράμμιση των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, τη εμπορική δηλαδή πολιτικής, της αλληλευτικής, τη κοινή αγροτική πολιτική, προκειμένου να επιδιωχθούν αναπτυξικοί στόχοι της Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει του άρθρου 208 της, Ευρωπαϊκής, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση των ε, επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής απόκρισης και της πρόληψης για τις φυσικές καταστροφές, κατά πολέμηση της διεθνούς ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, χρηματοδότηση της ανάπτυξης, μεταξύ, της, μεταξύ άλλων η επίσημη, η επίσημη κρατική παρέμβαση και ο έλεγχος των παράνομων ροών από, τις, από και προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μετά την ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί για την έκθεση του κυρίου Μίτσελ, για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, την ενδιάμεση αναθεώρηση του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξικής συνεργασίας και μετά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας και συντονιστής της ομάδας ε, Νίρ Σιντέβα, προτείνει στη δεύτερη προτεραιότητα να προσθεθεί η αναφορά στο σεβασμό των εξουσιών δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου. Συμφωνείτε? Μία τροποποίηση του κειμένου τελευταία στιγμής. Νομίζω ότι μόνο να ωφελήσει μπορεί μια τροποποιηση του κειμενου τελευταια στιγμή. νομιζω οτι αλλαγή. Οι συντονιστές επίσης ενέκριναν μια δομή για την διοργάνωση των ακροάσεων που θα λαμβάνει υπόψη τι εξή αρχέ. Ε, προκαταρτική ομιλία του προτινόμενου Επιτροπή για του Συντονιστέ. Ε, ισόρροπη κατανομή του χρονομιλία μεταξύ των ε, ε, ομάδων και ε, λήψη λόγου σε μορφή πινκ-πονγκ από τους εκπροσώπους των ομάδων και έπειτα απαντήσεις του προτινόμενου επιτρόπου. Η μερίση διάταξη των ερχόμενων συνεδριάσεων. Οι συντονιστέ θα εξετάσουν προτάσει και αιτήσει που μα υποβλήθηκαν για συζητήσει με άλλα θεσμικά όργανα και από οργανισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία. Νομική αποτίμηση. Αποφυνθήκαμε στην νομική υπηρεσία για γνωμοδότηση σε σχέση με τι συνέπειε από την υλοποίηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα την 1η Δεκεμβρίου για τη διασφάλιση και τη συνέχιση του άσκηση του δικαιώματο δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο και πώ αυτό θα υλοποιηθεί, θα κατά την εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαδικασία τη επιτροπολογία. Μελέτε. Θα αναθέσουμε μελέτη για την ενδεχόμενη μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να επιτρέψουμε στην τράπεζα αυτή να βελτιώσει τι συνθήκε δανειοδότηση ε, στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ζητήσαμε από τις υπηρεσίε μελέτης να κάνουν ένα απολογισμό των υπαρχουσών μελετών για την κερδοσκοπία και για τις πρώτες ύλες και κυρίως αυτές που απευθύνονται στην ανθρώπινη κατανάλωση, δηλαδή τα τρόφιμα. Αντιπροσωπίζεται το 2010 χρονοδιάγραμμα. Υιοθετήσαμε ένα χρονοδιάγραμμα για τι ακροασει των αντιπροσωπιών που αποφασίσαμε να ε, συγκαλέσουμε το 2010. Ενημερωτική συνεδρίαση για του βοηθού του Κοινοβουλίου. Αποφασίσαμε να είμαστε χορηγοί ως ε, Επιτροπή ανάπτυξη ε, των ε, συναντήσεων των ενημερωτικών που ενεργανώνται για του βοηθού του Κοινοβουλίου, όχι μόνο τη δική μα τη Επιτροπή, αλλά και άλλων επιτροπών όπω τη ΑΦΕΤ και τη ΙΝΤΑ. Τέλος, 17 Νοεμβρίου, τα μέλη της Concord οργανώνουν ε, μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία και εμείς θα είμαστε υποστηρικτές. Και τώρα, να δούμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε το 2008 να υιοθετήσει πρόσθετες κυρώσεις για τη Σομαλία. Αυτό που σήμερα συζητούμε είναι η υλοποίηση κάποιων τμήματων ε, των κυρώσεων σε σχέση με κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου επίσης. Πρόκειται για ένα ντοσχέ το οποίο θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον εισηγητή για να εξηγήσει τις τροπολογίες αυτές, να τις παρουσιάσει, καθώς και το που έχει φτάσει η όλη διαδικασία. Κύριε Φίλιπ Κάσμαρεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποιες επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές που θα προκύψουν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Εδώ μιλάμε για σοβαρές αλλαγές που μας περιμένουν. Η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να μας προσδώσει μια νέα νομική βάση, την, το άρθρο 215 της συνθήκης. Η κατάσταση είναι κάπως περίπλοκη, διότι γνωρίζουμε ότι ως τις 30 Νοεμβρίου το Συμβούλιο δεν θα έχει προλάβει να εγκρίνει τον κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όμως ήδη τη νέα νομική βάση. Η κατάσταση αυτή έχει επιπτώσει και στην έκθεση που ετοιμάζεται για τη Ζιμπάμπουε, η οποία θα συζητηθεί στο Στρασβούργο στην ερχόμενή μα συνεδρίαση. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό με το άρθρο 215 είναι το εξή. Πολύ συχνά λέμε ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα διευρύνει τι αρμοδιότητε του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό ισχύει μεν, αλλά εδώ έχουμε ένα από τα λιγοστά παραδείγματα, τι λιγοστέ περιπτώσει όπου τα πράγματα αντιστρέφονται. Εάν η επικεφαλής επιτροπή και η συνάδελφος Στρίφλερ είναι εδώ υπεύθυνη, εισηγήτρια, δεν μπορέσει να αποδεχτεί την έγκριση της έκθεσης ως την 1η Δεκεμβρίου, γιατί δεν θα υπάρχει νομική βάση, δεν θα υπάρξει και καμία πρόοδος. Η αρμόδια λοιπόν επιτροπή δεν θα εγκρίνει την έκθεση εγκαίρως. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή, η έκθεση δεν θα υπάρξει στην ουσία η διαδικασία αυτή βάσει της συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις διαβούλευσης με το Ευρωκοινοβούλιο. Συζητάμε το θέμα αυτό, συζητάμε διαφορετικές επιλογές που ίσως υπάρχουν, ποιες είναι οι ενδεχόμενες λύσεις, αλλά και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ νομίζω υπάρχουν παρόμοιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Προκειμένου να διατηρήσουμε την επιρροή του Ευρωκοινοβουλίου και προκειμένου να μπορούμε ακόμη να εκφράσουμε τις απόψεις μας, νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει απόφαση, απόφαση μετά τη συζήτησή μας. Θα έχουμε εδώ μια μεγάλη ευκαιρία η αρμόδια επιτροπή και η δική μας επιτροπή να αναλάβουν δράση, να εκφράσουμε την άποψή μας. Πάντως να προσθέσω εδώ ότι όλα αυτά σημαίνουν ότι θα έχουμε διαβουλεύσει σε προαιρετική βάση. Δηλαδή δεν θα υποχρεωθεί το Συμβούλιο να διαβουλευτεί με το Κοινοβούλιο τουλάχιστον δυνάμει τη συνθήκη. Οι διαβουλεύσει αυτέ θα είναι προαιρετικέ. Μπορούμε να προβάλλουμε και το επιχείρημα που θα λέει ότι εφόσον η συζήτηση για τον κορονισμό έχει ήδη ξεκινήσει βάσει τη συνθήκη τη Νίκαια, αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιπλέον δικαιώματα να περάσουμε σε προαιρετικές διαβουλεύσεις. Εάν η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ λοιπόν προωθήσει την πρόταση αυτή, πρόταση που αφορά, την, ε, που αφορά το προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο, θα πρέπει και εμείς να στηρίξουμε αυτή την ιδέα, διότι καθ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Τώρα επί το περιεχομένου, το ζήτημα των κυρώσεων είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω. Πρόκειται για ένα ζήτημα σοβαρό. Όχι μόνο για μα, αλλά για όλο το σώμα. Διότι εδώ μιλάμε για το βαθμό κατά τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι κυρώσει κατά των καθεστώτων, κατά των συστημάτων, όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη να επιβληθούν τέτοιε κυρώσει. Μια από αυτέ τι χώρε είναι η Σομαλία. Η Ζιμπάμπο είναι μια άλλη τέτοια περίπτωση. Η κατάσταση εδώ δεν είναι απλή, διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχει συντάξει κατάλογο για τα πρόσωπα τα οποία θα στοχεύουν οι κυρώσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν εμείς να ορίσουμε ποια είναι τα άτομα, τα πρόσωπα που εμείς θα, θέλουμε να στοχεύσουμε με αυτές τις κυρώσεις και ποια τα θεσμικά όργανα που θα φορούν οι κυρώσεις. Έχουμε αναφέρει κάποιες, κάποια από τα πρόσωπα αυτά. Μιλάμε για ανθρώπους που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, που διακινούν όπλα. Και ένα παράδειγμα αναφέρθηκε από τον κύριο Γκερέρο. Μιλάμε για ανθρώπους που κατέστησαν αδύνατη την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι στοχευμένες αυτές κυρώσεις θα οδηγήσουν στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, πάγωμα των θεωρήσεων. Και αυτό βεβαίω σχετίζεται και με το οικονομικό ζήτημα που προηγουμένω αναπτύξαμε. Η τελευταία αυτή κύρωση βρίσκεται στην, ε, ανάγεται στην αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Οπότε μόνον ε, με διαβούλευση με το κοινοβούλιο μπορεί να αποφασιστεί. Αυτά γενικά περί των κυρώσεων. Πάντω στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει γενικό συνένεση ότι οι στοχευμένε κυρώσεις κατά συγκεκριμένων προσώπων και φορέων ε, την κάνουν στήριξη. Εδώ, στην περίπτωση της Ομαλία, νομίζω ότι πρέπει να ε, υποστηρίξουμε και μέσα στοχευμένες κυρώσεις ή εκτός και αν δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα άτομα ή πρόσωπα. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νέες πληροφορίες για τη δράση, μάλλον για το έργο του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την έρευνα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα πρόσωπα αυτά και τα κατά πόσον θα επιβληθούν κυρώσεις. Οι τροπολογίες τώρα αφορούν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα την αποτελεσματικότητα, κάτι που συχνά συζητάμε. Προκειμένου οι κυρώσεις αυτές να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση, πιο τακτική αποτίμηση τέτοιου της επιβολής των κυρώσεων. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε αξιολογήσεις από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, τους οποίους θα μπορούσε να διορίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα έπρεπε να παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο. Δεύτερη τοπολογία, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι δεν πρέπει να παραβιάσουμε κάποιες προδιαγραφές, κάποια πρότυπα, κάποια δικαιώματα και να θυμόμαστε ότι ακόμη και όσοι, στοχεύουμε με τις κυρώσεις δεν πάβουν να έχουν κάποια δικαιώματα. Μπορεί να καταλήξουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των προσώπων που στοχεύουμε με τις κυρώσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα ανεξάρτητο κριτήριο κάλυψης των δικαιωμάτων των ανθρώπων ε, στους οποίους ε, θα, με τους, τους οποίους θα στοχεύουμε με τις κυρώσεις. Επίσης είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία αφαίρεσης ονομάτων από τον κατάλογο και εδώ το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται τακτικά και στη φάση της συμπερίληψης νέων ονομάτων στον κατάλογο, καθώς και τη φάση της αφαίρεσης των ονομάτων αυτών από τον κατάλογο. Σε κάθε περίπτωση το Κοινοβούλιο να λαμβάνει γνώση. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα να ακούσουμε αν γίνεται την ανάλυση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν, αν μπορείτε, να μα ενημερώσετε για τα όσα έγιναν στο Συμβούλιο τη ασφαλεία σε σχέση με αυτέ τι κυρώσει. Thank you, Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάξαμε την πρόταση μετά από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που χρονολογείται από έτους και βέβαια την εποχή της σύνταξής της δεν ήταν γνωστόν της πρότασης δηλαδή αν θα ε, κυρωθεί τελικά από όλες τις χώρες μέλη η συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπου πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Πώς θα πρέπει η πρόταση ή το σχέδιο κειμένου του Συμβουλίου να ενημερωθεί, να γίνει επίκαιρο. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, η μόνη νομική βάση που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη είναι το άρθρο 215 για τις προτάσεις που αναφέρονται στη Σομαλία και Ζιμπάμπουε. Εάν υπάρχει όμως και η πρόταση που αναφέρεται στις κυρώσεις κατά τα Λιμπάν και Κάιδα. Εάν αυτό εννοούσατε ε, με την ερώτησή σας περί νομικής ανάλυσης, η απάντησή μας είναι ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι το άρθρο 215 είναι ε, η σωστή νομική βάση και αντικαθιστά την νομική βάση τα, ε, αντικαθιστούν τα προηγούμενα άρθρα ε, της ε, ισχύουσας συνθήκης. Το 215 προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνουν από κοινού προτάσεις από τον ύπατο εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων και ε, πολιτικής ασφαλείας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι το νέο στη συνθήκη, εξ όσων γνωρίζω. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει η πρόβλεψη αυτή υπό, τις, ε, υπό τους παρόντες κανόνες. και ο εισηγητής μιλεί για την ανάγκη αξιολόγησης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην λησμονείτε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ Εθνών που βασίζονται στο άρθρο 7 του ε, καταστατικού των ΗΕ είναι δεσμευτικά για τις χώρες μέλη. Και γι' αυτό δεν είναι σύνηθες να γίνεται αξιολόγηση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κρίνει εάν το μέτρο θα πρέπει να παραμείνει ή να τροποποιηθεί. Το ψήφισμα προβλέπει ότι η αναθεώρηση αυτή πρέπει να ακολουθήσει μετά από ένα έτος. Άρα ήδη θα πρέπει να διεξάγεται σχετική συζήτηση στη Νέα Υόρκη. Και εάν οι κυρώσεις εφαρμοστούν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αυτόνομη βάση, θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαδικασία αναθεώρηση. Αλλά επειδή οι κυρώσει υπό το διεθνέ δίκαιο είναι δεσμευτικέ, ίσω να μην είναι σωστό να μιλούμε για την πρόταση που αφορά τη Σομαλία. Εν τέλει, δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κατάλογος προσώπων ή φυσικών ή νομικών οντοτήτων που να πλήττεται, να θίγονται από αυτή την, ε, κυρώσει από τη Νέα Υόρκη. Εάν ωστόσο αποδειχθεί αύριο ότι υπάρχει κατάλογος, ε, θα αναγκαστώ να παραδεχτώ ότι η Ένωση δεν μπορεί να, τον, ε, να τις εφαρμόσει τις κυρώσεις αυτές, διότι δεν υπάρχει σχετική διαδικασία. Δεν αποκλείεται το Συμβούλιο Ασφαλείας να περιμένει μέχρι ότου να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν εκδώσει τους καταλόγους αυτούς. Εάν επιμείνετε δείτε τους καταλόγους πρώτα, μπορεί αυτό να φέρει σε δυσκολίες τις χώρες μέλη μας, οι οποίες δεν διαθέτουν ακόμη την ε, κατάλληλη νομοθεσία. Εσείς κύριε Κάσμαν. Εγώ θα είμαι σύντομος, μιλώ εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Άκουσα τι είπε για τη νέα νομική βάση. Νομίζω όμως ότι όλες οι αλλαγές ε, των νομικών βάσεων θα γίνουν μέσα σε ένα καλάθι ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με το ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε πριν από την 1η Δεκεμβρίου διότι και αν ακόμη υπάρχει αλλαγή στην νομική βάση μέχρι τη στιγμή εκείνη πάντως θα έχουμε δηλώσει εμείς εδώ στην Επιτροπή μας τις πολιτικές μας προθέσεις και έχουμε μια θεμητή βάση για να το πράξουμε αυτό. Ορισμένες άλλες επιτροπές λένε ότι ένας κανονισμός που αναθεωρούμε θα πρέπει να μπει κάτω από τη νέα συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με το επιχείρημα ότι μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι βολεύει καλύτερα το κοινοβούλιο. Πρέπει να δεχθούμε τα προβλεπόμενα από τη συνθήκη. Για τον λόγο αυτό νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνουμε την θέση μας αυτή, έστω και αν δεν την εγκρίνει εν τέλει η Ολομέρεια. Διόλου δεν ενδιαφέρει αυτό. Μου φαίνεται και λίγο γελίο να μιλούμε για τον ύπατο εκπρόσωπο σαν έχουμε δήθεν και χαμηλότερους εκπροσώπους ή και μεσαίους εκπροσώπους. Όλοι οι εκπρόσωποι της Κομισιόν είναι high representatives. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον εκπρόσωπο εξωτερικών σχέσεων και εξωτερικής ασφάλειας. γνωρίζοντας ότι ο εκπρόσωπος εξωτερικών σχέσεων και πολιτικής ασφάλειας μπορεί να ε, ε, εργαστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ότι τα ε, μέτρα που προτείνει το Συμβούλιο Ασφαλείας ή που επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι δεσμευτικά και έχουμε και τροπολογία υπαριθμών ένα του εισηγητή που αν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά λέει ότι η Κομισιόν αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού. Και αυτό πράγματι αναμένουμε και αξιώνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράττει διαρκώ. Η εφαρμογή έχει γίνει σωστά. Αυτό μα ενδιαφέρει. Και αυτό μου φαίνεται να είναι ο σωστό τρόπο για να προχωρήσουμε. Και τώρα για τον εισηγητή. Μήπω είμαστε κάπω υπεραισιόδοξοι ζητώντα ετήσια βάση. Εγώ θα προτιμούσα βάση αναδιετία. Θα ήταν καλύτερο για να δούμε πώς λειτουργεί. και για να μην υπερεπιβαρύνουμε το προσωπικό της Κομισιόν, το οποίο δεν είναι και ε, πάρα πολύ πολύ αριθμό. Τώρα για την τροπολογία 2 που ε, προβλέπει προσθήκη στο ε, άρθρο 11 νέο και που λέει ότι τηρείται ενήμερο το Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε βήμα διαδικασία και για την τελική απόφαση. Για την τελική απόφαση το καταλαβαίνω, αλλά κάθε βήμα τη διαδικασία, όπω λέει το, εάν, ε, το άρθρο 11 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 είναι, είναι πράγματι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Μήπως πρέπει να δούμε καλύτερα τι θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Εσείς κυρία Στρίφλερ. Ευχαριστήσουμε τον Κάσμαρικ και την Γραμματεία της Επιτροπής Ελευθεριών είναι πολύ σύντομε οι προθεσμίε για τι τροπολογίε. Δηλαδή για την διαδικασία αυτή. Ε, ερωτήσεις με ψήφισμα. Για την Ζιμπάμπου επίσης, κύριος Μίτσελ, δεν θα σας πω ότι συμφωνώ μαζί του. Έκθεση για τη Ζιμπάμπου. Πρόεδρος. Ευχαριστώ από τώρα από πλευράς διαδικασίας έχω να σα προτείνω τα εξή. Η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών πρόκειται να λάβει την τελική τη οριστική απόφαση επί τη διαδικασία αύριο και πρέπει να προβλέψουμε τι εξελίξει για δύο διαφορετικά σενάρια. Στην απίθανη περίπτωση που αποφασίζει η Επιτροπή αυτή να εγκρίνει την έκθεση τέλο Νοεμβρίου, θα ε, κρατήσουμε ανοιχτό το θέμα και θα ψηφίσουμε 23 Ιανουαρίου. Σε αυτήν την περίπτωση η προθεσμία για τροπολογίε ε, καταλήγει αύριο 11 στι. στις το πιο πιθανό πάντως είναι η Επιτροπή Ελευθεριών να ζητήσει προφορική ερώτηση με ψήφισμα και για τη Σομαλία και για τη Ζιμπάμπουα. Στη αγγλική εκδοχή του κειμένου ε, έχει γίνει ότι χρειάζεται για να το λάβετε εσείς. Ο κ. Ε, Ντίβα επίσης για την ε, άλλη έκθεση είχε πει ότι πρόκειται να φροντίσει ούτως ώστε στην Επιτροπή Ελευθεριών να εμπλακούμε κι εμείς. 12 δεκάτου. Την Πέμπτη δηλαδή, η Επιτροπή Ελευθεριών πρόκειται να αποφασίσει, επομένως θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να εμπλακούμε στην προφορική ερώτηση. Πάντως, επίσημα πρόκειται να διαβιβάσουμε το κείμενό μας στην κυρίως αρμόδια επιτροπή μέχρι αύριο το απόγευμα. Και θα επιστρέψετε μια επιστολή όπου θα υπάρχουν κάποιε επεξηγήσει για τον προβληματισμό μα για το τι έγινε για την καθυστέρηση που σημειώθηκε σε σχέση με αυτά τα οποία αποφάσισαν με έγραφη διαδικασία οι συντονιστέ. Και να δούμε κατά πόσο να καταλήξουμε σε κάποιο σχέδιο κειμένου για ψήφισμα μαζί με την προφορική ερώτηση. Συμφωνείτε? Thank you. Then we will proceed. Πολύ ωραία. Τότε θα, σα προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ήταν προσταλή τον Μπαγκλαντές. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Μια από ο κύριος Ντίβα έχει υποχρέωση να βρίσκεται κάπου αλλού. Τώρα, ε, έχετε κάτι άλλο στα διάφορα. Όχι. Α, έχετε, έχετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα τα πω στα σου ειδικά με την αδειά σας. Ήθελα, επειδή έχω μιλήσει πολύ για συμφωνίες αλίας στην Επιτροπή αυτή και έχω μιλήσει και για συμφωνίες αλίας με, με χώρες τρίτου κόσμου και την πολιτική ανάπτυξη. Θέλω να σας ειδοποιήσω ότι έχω την 1η Δεκεμβρίου οργανώσει ένα δείπνο με συμμετοχή μιας σουηδικής οργάνωσης προστασίας της φύσης η οποία πρόκειται να υποβάλει μια έκθεση για το πώς θα πρέπει να διαρθρώνονται οι συμφωνίες αυτές ώστε να συμβαδίζουν με την πολιτική της ανάπτυξης και αυτό ήθελα να σας γνωστοποιήσω. Μάλιστα, η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στο Στρασβούργο στις 23 Νοεμβρίου Δευτέρα στις 7 το βράδυ μέχρι τις 8.30 και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από 8 μέχρι 11. Στις Βρυξέλλες θα είναι στις 10 Δεκεμβρίου, 5η, από 9 έως 12.30. Και με αυτό το μήνυμα